συμπεράσματα της συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17 η και 18ης Μαρτίου 16 και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Ντόναλτ Τουίσκ που έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχα πει τον Ιανουάριο εδώ στη Σύνοδο του Κοινοβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο δύο μήνες μπροστά της για να διασώσει τη ζώνη Σέγγεν και ότι στη Σύνοδο Συμβουλίου του Μαρτίου θα ήταν η τελευταία στιγμή για να δούμε αν έχει πετύχει η στρατηγική μας. Εάν δεν είχε επιτύχει, θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές επιπτώσεις, όπως η κατάρρευση του χώρου Σέγγεν. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε αυτούς τους μήνες. Ε, συγκάλεσα δύο συνόδους, οι οποίες αφοσιώθηκαν ακριβώς σε αυτό το θέμα, σχεδόν αποκλειστικά. Στις 7 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε τρεις σημαντικές αποφάσεις. Η πρώτη, ο τερματισμός της μέχρι τώρα προσέγγισης που σημαίνει ότι η ροή λαθρέων μεταναστών θα περνούν από τη Βαλκανική Οδό και θα φτάνουν εκεί που θέλουν. Αυτό έπαυσε. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην εικασία ότι η Ευρωπαϊκή Λύση δεν ε, γινόταν σεβαστή από την Ευρωπαϊκή δεν μπορούσε να, να συνταχθεί με την νομοθεσία, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις διατάξεις περί χώρου Σέγγεν. Η δεύτερη απόφαση είχε να κάνει με τη μαζική αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ελλάδα. θεσπίσαμε ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης με 3 εκατομμύρια, που θα 300, ε, εκατομμύρια ευρώ που θα σταλούν ήδη φέτος και ε, του χρόνου θα υπάρξει η συνέχεια ώστε να αντιμετωπιστούν οι τεράστιε συνέπειε τη άφηξη προσφύγων. Επίση, ειδική βοήθεια για να προσδεθούν τα εξωτερικά σύνορα στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και αυτά με την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία και την Αλβανία. Και άλλε μορφέ στήριξη εκφράστηκαν από τα κράτη-μέλη. Η τρίτη απόφαση αφορούσε τον επαναματρισμό προσφύγων, ε, μεταναστών μάλλον από την Ελλάδα στην Τουρκία, αυτών που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας. Καλωσορίσαμε την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για να ενισχύσει τις διαδικασίες ε, προστασίας και μυστικών υπηρεσιών, η Τουρκία συμφώνησε να, λάβει όλους να πάρει πίσω όλους τους μετανάστες που συλλαμβάνονται στα σύνορά της. Στο πρώτο αυτό συμβούλιο του Μαρτίου μου ζητήθηκε από τους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων να, υποβα... να εξετάσω τις προτάσεις της Τουρκίας και να καταλήξω σε μια κοινή ευρωπαϊκή θέση με σκοπό να φτάσουμε σε συμφωνία αργότερα μέσα στον μήνα Μάρτιο. Η συμφωνία αυτή τελικώς εξετάστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Μαρτίου. Συμφωνήσαμε όλοι οι παράτυποι μετανάστες που φτάνουν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά από τις 20 Μαρτίου και μετά θα επιστρέφονται στην Τουρκία. Η υλοποίηση θα, γινόταν, θα ξεκινούσε αμέσως και θα βασιζόταν στην αρχή ένας προς ένα όπως ονομάστηκε. Όλα αυτά άρχισαν να γίνονται πράξη. Ε, κατά με, τα δύο βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας ήταν πρώτον να εγγυηθούμε την συμμόρφωση με όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους εξασφαλίζοντας ότι ο καθένας μετανάστης που φτάνει στην Ευρώπη θα ε, είναι αντικείμενο ατομικής μεταχείρισης μεταξύ άλλων και με, την, με το σεβασμό του κανόνα για την ε, ε, αποφυγή των συλλογικών απελάσεων και του μη επαναπατρισμού. Ευχαριστούμε πολύ όλου και μεταξύ άλλων τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αφοσίωσή του και τη δουλειά του προ το στόχο αυτό. Έπειτα για τι ε, διαδημοκρατεύσει προσχώρηση. Ακούσαμε και τι κυπριακέ μέρημνε εδώ. Η προσέγγιση μα στο θέμα αυτό ήταν να τονίσουμε και να δούμε κατά πόσον μπορεί να σταθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προ όλα τα κράτη-μέλη. Και η Ευρώπη νομίζω ότι πέρασε αυτή τη δοκιμασία. Από την άλλη υπήρχαν πειρασμοί να πιεστεί η Κύπρος να κάνει τεράστιες παραχωρήσεις. Και αυτό είναι κατανοητό. Όμως από την αρχή παραμένα μετακίνητο στη θέση ότι δεν θα έπρεπε να θυσιάσουμε τα ε, ζωτικά συμφέροντα ενός κράτου μέλους, σε αυτή την περίπτωση της Κύπρου, στον βωμό της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. και κύριοι βουλευτές, γνωρίζουμε όλοι το τι υποχρεώσει και τι δυσκολίε έχουμε για να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε αυτή την κρίση. Τη εξ αρχή σκεφτόμουν ότι είναι επικίνδυνη πάτη να πιστεύουμε ότι υπάρχει ιδανική λύση που να είναι και 100% αποτελεσματική. Θέλω να πω σε όλους τους εκπροσώπου ε, και τους αναζητητές του πολιτικού Αγίου Δισκοπότηρου δεν θα το βρείτε ποτέ οι βολικές και τέλειες λύσεις δεν εξευρίσκονται στην, ε, στα πολιτικά πράγματα. Και σε αυτή την περίπτωση είναι και ανέφικτες. Αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι μια διαρκής και έντονη και ε, πολυδιάστατη προσπάθεια που πρέπει να καταλάβουμε, καταβάλουμε, η οποία δεν φαίνεται να φτάνει σε τέρμα. Οι λύσεις που εφαρμόζουμε μπορεί να μην είναι ιδανικές, αλλά ελπίζουμε να φέρουν κάποια αποτελέσματα. Και βεβαίως η ισορροπία που έχουμε εξεύρει δεν είναι τέλεια. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και κίνδυνοι και αδυναμίες. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βεβαιωθούμε ότι η συμφωνία ε, σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά παράλληλα είμαστε επιφυλακτικοί γιατί τα πάντα εξαρτώνται από το πώς θα υλοποιηθεί. Η συμφωνία με την Τουρκία και το κλείσιμο της Δυτικής Οδού των Βαλκανίων στέλνει ένα σαφέ μήνυμα προ την Τουρκία. Υπάρχουν και κάποιε αμφιβολίε προ τη χώρα αυτή και μερικέ από αυτέ τι συμμερίζομαι. Τι αμφιβολίε αυτέ μπορείτε να τι διασκεδάσουμε μόνον εάν οι λύσει εφαρμοστούν όπω συμφωνήθηκαν κατά και στην πράξη. Πρέπει επίση να λάβουμε υπόψη όλε τι αμφιβολίε και τι μέρημνε αυτέ και κάποιε να τι εκφράζουμε κιόλα. Να θυμίσω ότι ο βασικό στόχο που θεσπίσαμε ήταν να αποφύγουμε την λαθρομετανάστευση προς την Ευρώπη. Όπως έχω πει επανειλημμένως, χωρίς αυτό το στοιχείο και χωρίς την αποκατάσταση του ελέγχου της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης, δεν θα είμαστε σε θέση να προλάβουμε πολιτικές καταστροφικές συνθήκες. Εδώ εννοώ την κατάρρευση του χώρου Σέγγεν, την απώλεια ελέγχου των εξωτερικών μας συνόρων, με όλες τις συνέπειες που αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει για την ασφαλειά μας, το πολιτικό χάος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια, ε, μια κοινή αίσθηση ανασφάλειας και βεβαίως την ε, άνοδο του λαϊκισμού και του εξτρεμισμού. Σήμερα ο καθένας πλέον έχει κατανοήσει πόσο υψηλό είναι αυτό το διακύβευμα και πόσο συνεχίζει να είναι υψηλό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι συνθήκες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μην λειτουργήσουν προς όφελός μας. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι ο μόνος τρόπος να αναχαιτήσουμε τη λαθρομετανάστευση είναι να λύσουμε τα γενεσιολογικά αίτια τη κρίση αυτή. Δηλαδή να σταθεροποιήσουμε τον κόσμο γύρω μα, τι χώρε γύρω μα. Θέλω να το πω με σαφήνεια. Πολύ συχνά αυτό ακούγεται ω άλοθη για να μην κάνουμε τίποτε, να μην λάβουμε κανένα μέτρο εδώ στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι εν τέλει θα κατανοήσουμε ότι η Ευρώπη δεν έχει τα κλειδιά για όλες τις πόρτες στα χέρια της, ούτε μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα αυτού του κόσμου. Έχουμε ανησυχήσει τόσο πολύ ψάχνοντας ε, την λύση για να ε, επιλύσουμε τα προβλήματα των άλλων που δεν έχουμε ασχοληθεί με τα δικά μας προβλήματα. Η κρίση αυτή έδειξε εύλωτα ότι πρέπει να ανακτήσουμε το αίσθημα υπευθυνότητας και ευθύνης για τους αυτούς μας. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε όλο τον κόσμο γύρω μα. Στου δύο αυτού μήνε που συγκεντρωθήκαμε στο τι οφείλουμε να κάνουμε στη δική μα την αυλή, καταφέραμε να αποκομίσουμε κάποια αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα αυτά κατέστησαν εφικτά χωρί να αντιμετωπίσουμε αναγκαστικά τα γενεσιουργά αίτια τη μετανάστευση όπω ε, τον ε, λοιμό ε, και την πείνα στην ε, υποσαχάρια Σαχάρα, την, ε, τον πόλεμο στη Συρία και τη σταθεροποίηση περιοχών από τη Λιβύη στο Αφγανιστάν. Δεν μπορούμε να λύσουμε δια όλε αυτέ τι κρίσει. Όμω, φαίνεται ότι η ένταση στις σχέσεις μας με τη Ρωσία, ε, το τι γίνεται στον Αγκόρνο Καραμπάχ, η αντιμετώπιση της θερμοκρατίας σε πολλές περιοχές είναι στοιχεία τα που μπορούμε να επιδιώξουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε ταυτόχρονα. Πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει βεβαίως τα γενεσούργα αίτια της ε, μετανάστευσης και αυτό είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για όλη τη διεθνή κοινότητα. Οπότε θα ε, εργαστούμε σκληρά επί του προγραμματός μας να αντιμετωπίσουμε την κρίση της μετανάστευσης που θα υποβάλουμε στη σύνοδο του G7 στην Ιαπωνία και του G20 στην Κίνα με στόχο να αυξηθεί κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που έχουν πληγεί. Δηλαδή η αγορά εργασία, οι υποδομέ και οι εμπορικέ του ε, συνθήκε καθώ και ο κοινωνικό του ιστό. Να μην ξεχνάμε βεβαίω ότι να αντιμετωπίσουμε τα γενεσιουργά αίτια τη μετανάστευση θα είναι μια διαρκή μακροχρόνια προσπάθεια. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι ότι δεν θα έχουμε καμία εγγύηση ότι θα φτάσουμε σε απόλυτη επιτυχία. Διότι δεν εξαρτάται από τι δικέ μα δράσει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί πάνω απ' όλα εκεί όπου όλα εξαρτώνται αποκλειστικά από εμά. Δηλαδή το να διαχειριστούμε την κρίση στο ευρωπαϊκό έδαφος. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σε αυτό το πνεύμα πρέπει να ενεργήσουμε και να θυμόμαστε ότι η Βαλκανική οδός δεν είναι η μόνη. Και άλλες χώρες αναμένουν τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μας. Όχι μόνο η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Έχω κατά νου την ε, οδό της Κεντρικής Μεσογείου, εκεί που οι μετανάστες και από τη Λιβύη φτάνουν ε, σε βαθμό που ε, μπορεί να μας πραγματικά να μας ανησυχήσει. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αφήξεις στην Ιταλία. Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε ακριβώς τις λύσεις που εφαρμόσαμε στα Βαλκάνια, ακριβώς επειδή και η Λιβύη δεν είναι σταθερή ακόμα. Σε ό,τι αφορά τη Βαλκανική οδό, η δράση μας αναλήφθηκε πολύ καθυστερημένα. Και γι' αυτό υπήρξε και το προσωρινό κλείσιμο των συνόρων. Εντός της Ευρωζώνης πρέπει να συνεργαστούμε πλήρως με τη Μάλτα και την Ιταλία σήμερα προκειμένου αυτό το σενάριο να αποφευθεί και στο μέλλον. Κυρίε και κύριοι, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Ευρώπη ήταν διχασμένη. Υπήρχαν οι συνήγοροι της ασφάλειας και η υπέρμαχη του ανοιχτού πνεύματος. Σήμερα πρέπει επιτέλους να γεφυρώσουμε αυτές τις δύο διαφορετικές απόψεις, τις μεγάλες μας ανάγκες, ανάγκες για ασφάλεια στα σύνορά μας και την ανάγκη για να είμαστε ανοιχτοί και ανεκτικοί. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία των τελευταίων μηνών. Αυτή η συνθετική λύση θα είναι το μεγάλο, ε, το μεγάλο πεδίο μάχης για την Ευρώπη στο άμεσο μέλλον. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Σε αυτέ τι κρίσιμε στιγμέ τη ιστορία τη, η Ευρώπη υπήρξε νικηφόρα μόνον εφόσον ανέλαβε την ευθύνη και ε, αντιμετώπισε αυτέ τι δυσκολίε ταυτόχρονα. Ω πραγματικοί Ευρωπαίοι πρέπει να παραμένουμε ανοιχτοί και ανεκτικοί, αλλά ταυτόχρονα και να επιδείξουμε πυγμή και, και αποτελεσματικότητα. Οι εντάσει είναι αναπόφευκτε. Η ευρωπαϊκή δεξιότητα ήταν να τις μεταλλάξει σε θετική ενέργεια και αυτήν μας την τάση πρέπει να τη διατηρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τουίσκ. Και τώρα το λόγο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο πρόεδρος κύριος Γιούγκερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές. η βία των φανατικών, η τυφλή βία, αυτό είναι αυτό που γνωρίζουν καθημερινά ε, πολλές χιλιάδες πρόσφυγες στη Συρία και αλλού και προσπαθούν να ξεφύγουν. Προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη, πολύ συχνά πέφτουν στα χέρια διακινητών, οι οποίοι αγοράζουν φτηνά σκάφη ε, με πολύ φτηνή τιμή καταφέρνουν να έχουν τεράστια έσοδα, εκτιμώντας τα 3 με 6 δις ευρώ το 2015. Αυτήν την ε, ανθρώπινη δυστυχία προσπαθούμε να την αντικαταστήσουμε με ε, μετακίνηση πληθυσμών συμφωνημένη. Αυτό είναι ο στόχο τη συμφωνία, στην οποία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία 18 Μαρτίου. Αυτή τη συμφωνία αρχίσαμε να εφαρμόζουμε. Είτε θα δεχθείτε ότι το νόμο στο Αιγαίο τον κάνουν οι διακινητές και οι εγκληματίες είτε θα δεχθείτε ότι έχει έννοια η προσπάθεια αυτή που κάνουμε αυτή η συμφωνία που προσπαθεί να ρυθμίσει τις ε, προσφυγικές ροές μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά δεν είναι εύκολο. Απ' την αρχή το είπα. Θα είναι Ηράκλειος άθλος και είναι η εφαρμογή είναι ευθύνη των ελληνικών αρχών και των τουρκικών αρχών. Αλλά η επιτυχία αυτής της συμφωνίας είναι η κοινή μας ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιτόπου με το συντονιστή της τον κύριο Μάρτιν Βερβέ που συνεργάζεται σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τις ελληνικές αρχές, τις τουρκικές αρχές για να τους βοηθήσει στην εφαρμογή, στην πράξη αυτής της συμφωνίας προσέχοντας την ουσία δηλαδή τον πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Από τις 4 Απριλίου, όταν άρχισε να ισχύει αυτή η συμφωνία, μέχρι σήμερα 325 παράτυποι μετανάστες έχουν επιστραφεί από την Ελλάδα στην Τουρκία και 79 Σύριοι πρόσφυγες μετεγκαταστάθησαν από την Τουρκία στην Ευρώπη. Είναι μόνο η αρχή. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία, όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για να λειτουργήσει αυτό το καθεστώς και επιστροφών και μετεκαταστάσεων. Η ευθύνη μας για τους ε, πρόσφυγες, κύριε Πρόεδρε, δεν σταματά στα εξωτερικά σύνορα. Σημεία αφετηρίας του σχεδίου δράσης με την Τουρκία είναι να δράσουμε από κοινού ούτως ώστε να υπάρξουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και προοπτικές για τους πρόσφυγες. Γι' αυτό τα τρία δις που εγκρίναμε είναι πολύ σημαντικό ποσό και είναι σωστό και σημαντικό μέχρι τέλος του 18 να παράσχουμε άλλα τρία δις. Διότι τα ποσά αυτά δεν θα παρασχεθούν στην Τουρκία όπως ε, συχνά διαβάζω. Αυτά τα ποσά, αυτές οι πιστώσεις θα διατεθούν για τους πρόσφυγες ούτως ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες τους, τις ανάγκες στέγασης, τις, τις ανάγκες ε, διατροφής, τις ανάγκες εκπαίδευσης για τα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά τους έχουν δικαίωμα να έχουν προοπτική μέλλοντος. Και ήδη είμαστε σε φάση εκπόνησης ε, των αναγκαίων διατυπώσεων για να παρασχεθούν τα πρώτα ποσά. Και έχουμε δώσει ήδη την εντολή να ε, διατεθούν 55 εκατομμύρια για να δώσουμε σχολική εκπαίδευση και άλλα 40 εκατομμύρια θα δοθούν για διατροφική βοήθεια από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και με αυτόν τον τρόπο πολλές χιλιάδες σύρων προσφύγων θα μπορέσουν να λάβουν την αναγκαία διατροφή και άλλα προγράμματα είναι υπό προετοιμασία ή υπό εφαρμογή. Συχνά τίθεται το ερώτημα και εδώ εάν η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος. Και δεν θέλω ε, να αποφύγω να πω ότι υπάρχουν διάφορα θέματα επί των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία έχουν εντελώς διαφορετικές ε, απόψεις. Αλλά είναι σαφές επίσης το εξής. Επειδή εκτιμούμε ιδιαίτερα η προσπάθεια εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσπάθεια που πρέπει να γίνει από όλου για την ε, βοήθεια στους πρόσφυγες αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα εκφράσουμε τη διαφωνία μας για τα θέματα που υπάρχουν στην Τουρκία, για παράδειγμα για τα θέματα του, της ελευθερίας του τύπου. Δεν καταλαβαίνουμε πώς είναι δυνατόν να καλείται ο Γερμανός πρέσβης για να δώσει εξηγήσει για ένα δημοσίευμα το οποίο μπορεί να είναι αυθάδες. Αυτό δεν μας βοηθάει να υπάρξει προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά αντίθετα μας απομακρύνει. Η εταιρική σχέση με την Τουρκία όμως μας δίνει και κάποιες τέτοιες δυνατότητες γιατί μέσω του διαλόγου μπορούμε να συζητήσουμε τα βασικά θέματα που μας ενδιαφέρουν και ελπίζουμε να ενδιαφέρουν και την Τουρκία. Μας επιτρέπουν να τα συζητήσουμε πιο εκ του σύνεγγης και εάν η Τουρκία μέσω των διαπραγματεύσεων ένταξης προσεγγίσει τις θέσεις μας τότε δεν μπορώ παρά να το χαιρετήσω αυτό και ελπίζω, ελπίζω να μπορέσω να τη χαιρετήσω και εντός ε, ε, της Ένωσης κάποια στιγμή. Η συνεργασία ε, πρέπει να είναι και από τις δύο πλευρές. Και μπορούμε να βοηθήσουμε μόνο αν συνεργαστούμε πολύ πιο στενά. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το εξής επιπλέον γεγονός. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί σχεδόν 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα και περισσότερα από όσα έχει υποδεχθεί όλη η Ευρώπη. Άρα δεν πρέπει να αφήσουμε μόνη της την Τουρκία με αυτή την ευθύνη. Αυτό είναι θέμα αλληλεγγύης. Βεβαίω, εφόσον μεταξύ μα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, τότε πρέπει να υπάρχει και αλληλεγγύη έναντι εκείνων που έχουν αναλάβει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Η αλληλεγγύη, κύριε Πρόεδρε, είναι ε, η κατευθυντήριά μα γραμμή στην προσπάθεια να αναθεωρήσουμε το κοινό σύστημα ασύλου στην Ευρώπη. Ξέρουμε τις αδυναμίες του τρέχοντος συστήματος και τις ξέρουν και οι διακινητές και έχουν εκμεταλλευτεί τις διαφορές των εθνικών νομοθεσιών για να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα τις αναλλακτικές λύσεις για μεταρρύθμιση του συστήματος. Τρία πρέπει να κάνουμε πιστεύω πάνω απ' όλα. Πρώτον, πρέπει να καταστεί σαφές ποιο κράτος μέλος είναι αρμόδιο για την ε, διαχείριση μιας αίτησης ασύλου. Αυτή είναι η βάση του κοινού συστήματος. Πρέπει να είναι σαφές, πρέπει να είναι εφικτό, πρέπει να είναι βιώσιμο ακόμη και σε περίοδους κρίσης. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά και παιδιά λαμβάνουν ε, βοήθεια με συνθήκες ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας όπου και αν είναι. Και τρίτον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο που αιτείται άσυλο θα διαμένει στη χώρα που έχει καθοριστεί ότι θα πρέπει να διαμένει. Είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των προσφύγων αλλά και την τήρηση των υποχρεώσεών τους από αυτούς. Αλλά ένα στοιχείο θα πρέπει να είναι η βάση οποιασδήποτε μεταρρύθμισης, η αλληλεγγύη. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του μία κρίση. Η θέση μιας χώρας ε, στο γεωγραφικό χάρτη δεν θα πρέπει να αποφασίζει πόσο βάρος θα πρέπει να φέρει. Θέλω να με βοηθήσετε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Έχετε δυνατότητα να μας δώσετε καθημερινές γραμμές πριν δημοσιεύσουμε τις προτάσεις μας τον επόμενο μήνα. Σας καλώ σήμερα να συμμεριστείτε τις ιδέες σας μαζί μας. Είμαι πολύ ικανοποιημένο που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18 Μαρτίου ενέκρινε την ε, στρατηγική της πολιτικής για την ε, ανάπτυξη και την απασχόληση. Θέλουμε να υπάρξουν και επενδύσεις και με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση. Αυτή τη στρατηγική θα εφαρμόσουμε, την έχουμε ήδη εφαρμόσει και έχει ήδη φέρει τα πρώτα αποτελέσματα η θέση στον κόσμο, η οικονομική θέση στον κόσμο εξακολουθεί να είναι λεπτή και η ανάπτυξη είναι ανεπαρκής και εξακολουθούμε να έχουμε 22 εκατομμύρια ανέργους και όσο έχουμε 22 εκατομμύρια συμπολίτες χωρίς εργασία δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει λήξει η κρίση. Μια μέρα πριν τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Κομισιόν καθόρισε τη στρατηγική της για τη χαλιβουργία. Και θέλω να κάνω έκκληση έντονη να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα προβλήματα της ευρωπαϊκής χαλιβουργίας, γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε βιομηχανία. Η χαλιβουργία έχει σταματήσει να είναι βαριά βιομηχανία. Η χαλιβουργία είναι ο τόπος, ο χώρος όπου εφαρμόζονται τεχνολογίες εχμής και οι χαλιβουργοί δεν είναι πλέον ανειδίκευτοι. Είναι εξαιρετικά ειδικευμένοι εργαζόμενοι. Και αυτοί οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι πρέπει οπωσδήποτε να στηριχτούν ανεπιφύλακτα. Το αξίζουν. Γι' αυτό πρέπει με κάθε αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της παγκόσμιας υπερπαραγωγής χάλιβα. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν στις τεχνολογίες μέλλοντος και στο προσωπικό που εργάζεται στον κλάδο αυτό. Στην Ευρώπη έχουμε 360.000 εργαζόμενους στη χαλιβουργία, αλλά αυτοί που έμεσα σχετίζονται με τον κλάδο είναι πολύ περισσότεροι. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτές τις θέσεις εργασίας. Αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα της ε, βιομηχανικής μας πολιτικής. Κύριε Πρόεδρε, το ελεύθερο εμπόριο πρέπει να είναι και δίκαιο εμπόριο. Αυτή τη στιγμή κάνουμε έρευνες για να δούμε εάν κινέζικα προϊόντα χαλιβουργία είναι αντικείμενο dumping και θα πάρουμε και άλλα μέτρα αν χρειάζεται. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον γεωργικό τομέα είναι σημαντική διάσταση του κοινού μας εγχειρήματο. Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πρόγραμμα δράσης για τον ΦΠΑ δίνοντας στα κράτη-μέλη περισσότερη ευελιξία για να καθορίζουν τους συντελεστές ανάλογα με τις προτεραιότητές τους. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σε εποχές αναταραχών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και να προωθεί λύσεις και να οικοδομεί γέφυρες. Αυτή είναι η αποστολή μας. Να υπάρξει σταθερότητα και θα συνεχίσουμε το έργο μας αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γιούνκερ. Εκ μέρους της ομάδας του ΕΛΚ, ο πρόεδρος κύριος Βέμπα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, επί μήνες συνδυάζουμε και ασκούμε κριτική κατά του Συμβουλίου ε, για την έλλειψη ενότητας. Ε, πρέπει να πούμε τώρα ότι στη συνεδρίαση πριν από το Πάσχα κατάφεραν να επιτύχουν μια, μια κοινή οδό για την Τουρκία και για μια λύση για το μεταναστευτικό κατάφερε η Ευρώπη, η αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να βρουν μια κοινή λύση και θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κ. Ντόναλτ Τούσκ, γιατί αυτό είναι το έργο του και κατάφερε να βρει ένα κοινό δρόμο στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, την απάντηση τη βρήκαμε μαζί με την Τουρκία. Υπάρχει μόνο ένα κοινό δρόμο η Τουρκία ήδη έχει σχεδόν 3 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στη χώρα και σεβόμαστε αυτή την προσπάθεια. Λειτουργεί τώρα και το σύστημα που αποφασίσαμε για την επιστροφή των παρατύπων μεταναστών. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα συστήματα των διακινητών και προσπαθούμε να επαναφέρουμε την τάξη στο μεταναστευτικό και αυτό το οποίο ε, κάνουμε για την οδό των Βαλκανίων θα πρέπει να το κάνουμε και για την οδό της Μεσογείου όπως είπατε κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν θέματα τα οποία ε, θεωρούνται ε, παράτυπα κατά του κράτους δικαίου. Αυτό ισχυρίζονται οι κομμουνιστές και ο κύριος Τσίπρας πολλές φορές έχει ισχυριστεί Μερικές φορές όταν η αριστερά ασκεί κριτική θα πρέπει πολλές φορές να θέσει αυτά τα ερωτήματα και στην Ελλάδα. Και ο κύριος Φερχόφστατ για τον συνάδελφό του κύριο Ρούτε ως πρόεδρο του Συμβουλίου, του Συμβουλίου θα πρέπει να θέσουν τα, τα ερωτήματα αυτά στους, στις πολιτικές τους ομάδες. Η Ευρώπη χρειάζεται ασφαλή σύνορα, αλλά η Ευρώπη δεν είναι φρούριο χρειαζόμαστε νόμιμη οδό προ την Ευρώπη, ώστε άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη να μπορούν να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη και υποστηρίζουμε αυτές τις κινήσεις. Τους τελευταίους μήνες εκατοντάδες χιλιάδες πέρασαν χωρίς έλεγχο, χωρίς καταγραφή, χωρίς έλεγχο ασφάλειας και σύμφωνα με τις ε, ε, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις αποφάσεις της Μακεδονίας δόθηκε ένα τέλος ε, σε αυτή την εισρωή. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο είπε και ο Ζων Κλοντιούν και σήμερα. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να δώσουμε μια νέα αρχή στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Έχουμε μια εταιρική σχέση που φαίνεται ότι λειτουργεί και μπορούν οι δύο λαοί να ε, λειτουργήσουν από κοινού. να ξεκινήσει μια νέα πορεία με τον πρόεδρο Ερντογάν και εκείνο ε, να σέβεται τα δικαιώματα των ε, μειονοτήτων, τα δικαιώματα τη ελευθερία του τύπου. Διαφορετικά θα δείξει ότι δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει Ευρώπη. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την ελευθερία του τύπου ε, στην Τουρκία, αλλά ισχύει και για την ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο σεβόμαστε εμείς θέλουμε να σέβεται και ο πρόεδρος Ερντογάν, να σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες. Το δεύτερο θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν το θέμα της ανάπτυξης, αγαπητοί συνάδελφοι, και θα ήθελα και αυτό να το σχολιάσω. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη βλέπουμε θετικά αποτελέσματα. Χθε είχαμε τον ε, ε, πρόεδρο του ε, κόμματος του ΕΛΚ στην ε, ε, Κύπρο, στην ε, ομάδα μας στο ΕΛΚ γιατί η Κύπρος είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι κατάφερε να περάσει από το μνημόνιο στην ανάπτυξη. Με τις σωστές μεταρρυθμίσεις και με την σταθεροποίηση του προπολογισμού κατάφεραν να περάσουν σε κατάσταση ανάπτυξης αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ε, όταν ε, προς τους ψηφοφόρους πρέπει να λέμε ότι ε, οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να μπορούν να υπάρχουν και τα αντίστοιχα χρήματα. Είναι διδάγματα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Μην πιστεύετε αυτούς οι οποίοι υπόσχονται, όπως ο κύριος Τσίπρας, πολλά χωρίς να κάνει μεταρρυθμίσεις στη χώρα του. δεν μπορούμε να έχουμε τέλος των μεταρρυθμίσεων και μόνο να ζητάμε χρήματα. Πρέπει να εφαρμόσουμε μεταρρυθμίσεις, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τις χώρες μας, να έχουμε σταθερό προϋπολογισμό και αυτή είναι η γραμμή πάνω στην οποία κινείται η ομάδα του ΕΛΚ και θα συνεχίσει να κινείται. Ευχαριστώ πολύ. Äh, ο κύριος Λάμπερς θέλει κάνει μια ερώτηση. παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μάνφρεντ, αναφέρθηκες στο ότι ο κύριος Ερντοάν πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα τέτοια. Μα τι δυνατότητες πίεσης έχετε εσύ και η καγκελάριό σου. Δέχεστε ό,τι και να σας πει, μόνο για να κρατήσει τους πρόσφυγες. Ένας ε, κομικός στη Γερμανία κοροϊδεύει την κατάσταση και λέει ακριβώς ότι η καγκελάριος θέλει να ευχαριστήσει τον Ερντογάν και δεν ξέρει τι να πρωτοκάνει. Αν ήμουν ο Ερντογάν θα γέλαγα με αυτά που ακούω. Παρακαλώ, μπορεί να πει ο Ερντοάν, α πει ό,τι θέλει ο Μάνφρετ Βέμπερ, εγώ θα πω στην Καγκελάριο να μου κάνει όλα μου τα χατήρια και θα τα κάνει. Ο κύριο Βέμπερ, βλέπω ότι σα ε, χειροκροτεί η δεξιά για αυτά που λέτε. Συγχαρητήρια. Κοιτάξτε, ίσως να μην το γνωρίζουν ήδη οι πράσινοι, αλλά δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου της καγκελαρίου μου, εκπρόσωπος ε, και πρόεδρος του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να το καταλάβετε. Κοιτάξτε, σε κανένα δεν υποκλεινόμεθα για το θέμα των θεωρήσεων για παράδειγμα. Δεν θα υπάρξει ε, καμία παραχώρηση. Είτε η Άγκυρα θα εφαρμόσει όλα όσα απαιτούνται Αλλιώς δεν πρόκειται να τους ε, χορηγήσουμε ε, την ε, ελάφρυση των θεωρήσεων. Δεν κάνουμε κανένα παζάρι. Θα δείτε το κοινό ψήφισμα για την Τουρκία που θα ψηφίσουμε σήμερα, όπου το Κοινοβούλιο καθιστά σαφές ότι δουλεύουμε πραγματιστικά για να επιδιώξουμε κοινέ λύσεις με τους γειτονές μας, όποιοι και να είναι, αλλά παράλληλα λέμε ότι περιμένουμε να εφαρμοστεί το δίκαιο από την Τουρκία. Ελπίζω αυτό να ισχύσει ως στάση για όλα τα κόμματα. Και τώρα λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Πιτέλα για τους Ελληνοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα τα λόγια του Πρόεδρου Τούσκ. Η συμφωνία αυτή δεν είναι τέλεια, είπε. Και κατανοώ την αξιέπαινη και θετική πρόθεση του Πρόεδρου Γιούνκερ. Πρέπει να πάρουμε το μπαλάκι από τα χέρια των εμπόρων του θανάτου. Βεβαίως παραμένουν εμφιβολίες της ε, πολιτικής μου ομάδας. Έχουμε συνάψει συμφωνία. Στην στιγμή ακριβώς αυτή που η Τουρκία κλείνεται στα όρια της. Η ελευθεροτυπία καταπιέζεται και καταπατώνται τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Θα ζητούσα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο και να είναι σε επιφύλακη και να απαιτούν το σεβασμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο περί ανθρωπιστικών ε, συνθήκων στην Τουρκία. Η οικονομική στήριξη και οι ανθρώπινοι πόροι οφείλονται προς την Ελλάδα και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και τα παιδιά. Θα πρέπει επίσης να δούμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα ευρωπαϊκής διαχείρισης των hotspot. Με όλα αυτά θα πρέπει να πούμε μεταξύ μας το εξής ειλικρινώς. Επικρίνουμε αυτή τη συμφωνία και εγώ αυτό κάνω. Ωστόσο, αυτή τη συμφωνία υποχρεωθήκαμε από, τις, ε, από τον εγωισμό και την στενοκεφαλιά κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τη δεχτούμε, διότι αρνήθηκαν να έχουν επαναγκατάσταση, να δεχτούν την επαναγκατάσταση των προσφύγων. Κανείς από εμά δεν έχει στα χέρια του το μαγικό ραβδάκι για να επιλύει τα θέματα αυτά. Ξέρουμε όμω όλοι ότι το κλειδί για να κερδίσουμε αυτό το στίχημα είναι να έχουμε έναν υποχρεωτικό και αυτόματο μηχανισμό όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Και πρέπει να σκεφτούμε και την ιδέα επιβολής κυρώσεων κατά των χωρών που βάζουν τρικλοποδιά στο σύστημα. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε η Ένωση από τη μια να επιχρώνει ένα κράτος με 1,0% ε, έλλειμμα να να αναλάβει οικονομικές ε, υποχρεώσεις και να μην ε, στηρίζει τις επιχειρήσεις διάσωσης, να μην έχει μια σαφή πολιτική μετανάστευσης. Δεν μπορεί να είμαστε αυστηροί μόνο στους λογαριασμούς και να μην δίνουμε καμία σημασία στους ανθρώπους. Ε, μια τέτοια στρατηγική χρειαζόμαστε. Αλλά δεν είναι μόνο το πρόβλημα τα Βαλκάνια. Υπάρχουν σκάφη που φτάνουν διαρκώ στι νότιε όχθε μα και θα πρέπει να έχουμε και με τι αφρικανικέ χώρε ένα σύμφωνο για την ανάπτυξή του. Θα έχουμε μια νέα έξοδο του ερχόμενου μήνε προ την Μεσόγειο. Μετανάστε θα έρχονται από την Αφρική και από την Αλβανία. Και εμεί τι θα κάνουμε, θα χτίζουμε τείχη στο νερό τη θάλασσα. Το να πιστεύουμε ότι μπορούμε να σταματήσουμε με τύχη την άφηξη των ανθρώπων δεν είναι απλώς μη ρεαλιστικό, είναι σχεδόν επονίδιστο. Δείτε τι γίνεται στην Αυστρία. Τι είναι αυτό το προληπτικό τείχος για 25 μετανάστες ημερησίως, τι θα πει. Είναι άχρηστο, είναι και ντροπή και είναι και επιζήμιο. Τις ερχόμενες λοιπόν εβδομάδες έχουμε μια ιστορική ευκαιρία έχουμε την ευκαιρία που μας δίδεται από την δυνατότητα να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό του Δουβλίνου. Ο κύριος Γιούνκερ πρόσφερε ξανά ένα σύμφωνο συνασπισμό με το Κοινοβούλιο. Και εγώ λέω ναι. Λέω ναι στον πρόεδρο Γιούγκερ. Ναι, συμμαχία με το Κοινοβούλιο, αλλά με πραγματική και τολμηρή μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, που να πάει στην ουσία των κανόνων του Δουβλίνου και πραγματικά να θεσπίσουμε μια κοινή ε, πολιτική του ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, Πρόεδρε, και κλείνω, πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτά που μας ενώνουν. Οι φιλευρωπαϊκές δυνάμεις μας ενώνουν και βρίσκονται εδώ, στην Ευρώπη. Και να μην κοιτάζουμε αυτά που μας διαιρούν σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές. Ας αποφύγουμε να μετατρέψουμε αυτήν την σύνοδο ολομέλειας σε αρένα για τις εκλογικές μας εκστρατείες στην Ισπανία, την Ελλάδα, σε άλλες χώρες. Ας γίνει αυτό στις χώρες μας. Εδώ ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ενότητά μας και να κοιτάξουμε να αλλάξουμε και να σώσουμε την Ευρώπη. Πιτέλα, ο κύριο Ζούλικ θέλει να σα κάνει μια ερώτηση. Τη δέχεστε, παρακαλώ, κύριε Ζούλικ. Κύριε Πιτέλα, θέλετε να υπάρξουν κυρώσεις για τις χώρες που δεν δέχονται μετανάστες. Η ερώτησή μου είναι η εξής εάν ε, η ευρύτατη πλειοψηφία ε, των πολιτών μιας χώρας δεν θέλουν να δεχθούν εκατοντάδες χιλιάδες ε, μετανάστες πρέπει να αγνοήσουμε την άποψη των λαών αυτών παρακαλώ να μου δώσετε μια ε, απευθείας απάντηση εντελώ απευθεία, ούτε καν άμεση απάντηση. Εάν μια χώρα αποφασίζει ελεύθερα να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούται να συμμορφωθεί με τι αποφάσει που λαμβάνονται στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για το ECR ο κύριος Καμάλ. Το Σεπτέμβριο ο Φρανς Τίμερμαν στην Ολομέλεια μίλησε για, το, για την κρίση του προσφυγικού ε, και ε, μας είπε ότι είναι δραματική η κατάσταση όταν πλησιάζει ο χειμώνα. Ε, τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης εκτιμά ότι οκταπλάσια αριθμοί ατόμων ήρθαν το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το 2015. Ξεπεράσαμε τους αριθμούς των ε, προηγουμένων ε, μηνών και του καλοκαιριού. Κατανοούμε ότι προσπαθούν να ζητήσουν μια καλύτερη ε, ζωή στη χώρα μας και κανείς, δεν θέλει, κανείς μας δεν θέλει να χάνουμε χρόνο για να βελτιώσουμε και την αξιοπιστία των θεσμικών μας οργάνων και να μην επιβαρύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ανώφελα το καλοκαίρι που μας έρχεται θα έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε ότι μάθαμε αυτά τα διδάγματα τα οποία πρέπει να διδαχθούμε από το καλοκαίρι του 2015. Είπε ο κύριος Στούσκο ότι δεν είναι όλες οι συμφωνίες τέλειες. Πολλά έχουν γίνει για να αντιμετωπιστεί η κρίση και η ομάδα μας υποστηρίζει πολλές από αυτές τις αποφάσεις. Διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων, βελτίωση ε, της ζώνης Σέγγεν, βελτίωση του προγράμματος επανεισδοχής, ε, ε, αναχέτηση των διακινητών. Με αυτά συμφωνούμε. Υπάρχουν όμω και άλλε αποφάσει που μπορεί να μα κάνουν να νιώθουμε καλύτερα τώρα, αλλά μπορεί να δημιουργούν τεράστια προβλήματα για το μέλλον. Θαυμάζω βέβαια τον τρόπο με τον οποίο το τουρκικό έθνο ε, έχει 2,7 εκατομμύρια πρόσφυγε. και όπω είπε ο κύριο Τούσκ, πολλοί από εμά έχουμε ακόμη πολλέ αμφιβολίε για την ε, συμφωνία με την Τουρκία σε πρακτικό επίπεδο και σε νομικό επίπεδο και σε ηθικό επίπεδο και διοντολογικό επίπεδο και ο χρόνο θα δείξει τι θα γίνει με τη συμφωνία με την την Τουρκία. Μπορεί ε, η Γερμανή καγκελάριος να χαίρεται και τη συμφωνία με την Τουρκία, αλλά άλλες χώρες ε, θέτουν ε, πολλά ερωτήματα και πολλές ανησυχίες. Ζούμε σε μια εποχή των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και καταλαβαίνουμε ότι μόλις ένα σημείο ανοίξει θα κατακλειστούν τα κοινωνικά μέσα και θα, θα μάθουν όλοι από πού μπορούν να περάσουν, από την Ιταλία, από τη Μάλτα, από οπουδήποτε αλλού. Σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Δουβλίνου, βλέπουμε εναλλακτικέ λύσεις για τη μεταρρύθμιση. Μία εναλλακτική λύση είναι ότι ε, ο κανονισμός για το άσυλο αποτελεί ε, το ε, βασικό μέσο. Η δεύτερη λύση, η δεύτερη εναλλακτική είναι να λειτουργήσει καλύτερα ο κανονισμός που ήδη έχουμε. Υπάρχει τώρα επιλογή μεταξύ μια στρατηγική που είναι ιδεαλιστική με μικρές πιθανότητες επιτυχίας και μια στρατηγική που είναι ρεαλιστική και βελτιώνει την τρέχουσα κατάσταση. Νομίζω ότι οι πολίτες μας θα προτιμούν το ρεαλιστικό τη ρεαλιστική λύση και όχι τον ιδεαλισμό. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τους κανόνες που έχουμε να λειτουργήσουν σωστά και να μην αναζητούμε το χρυσό κλειδί που είπε ο κύριος Τούσκο θα άνοιγε όλες τις πόρτες. Ας καταβάλουμε προσπάθεια και ας δαπανίσουμε χρήματα για τον έλεγχο των συνόρων μας, να επιστρέφουμε τους ε, ε, μετανάστες που δεν ε, τους απειλεί ε, κίνδυνο της ζωή του, ε, να βελτιώσουμε τι εφιστάμενε τις εφιστάμενες ε, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ασύλου και να προσπαθήσουμε να εγκαθιστούμε πρόσφυγες ώστε να τον πιο κοντά στην πατρίδα τους και όχι σε περιοχές όπου θα κινδυνεύουν. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πολιτική ασύλου δίκαιη και σωστή που θα βασίζεται στον πραγματισμό και στην, στο ανοιχτό μας πνεύμα προς τους άλλους. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι απλό. Έρχεται το καλοκαίρι και δεν έχουμε χρόνο να επανεφεύρουμε τον τροχό. Έχουμε όμως χρόνο για να βελτιώσουμε το σύστημά μας. Κύριε Καμάλ, ε, ο κύριος Γκραπίνη, κυρία Γκραπίνη, θα ήθελε να σας κάνει μία ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Γκραπίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Καμάλ, είπατε επανειλημμένος ότι πρέπει να είμαστε πραγματιστές, ότι πρέπει να έχουμε νέα μέτρα ρεαλιστικά και να επιδείξουμε αλληλεγγύη και ανθρωπισμό. Εάν εσείς είσαστε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εσείς τι θα κάνατε. Πώς θα τα υλοποιούσατε όλα αυτά που λέτε ότι πρέπει να γίνουν. Γιατί μια ζωή μας λέτε τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν μας λέτε πώς. Τι θα κάνατε λοιπόν, αν είσαστε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπω ότι με κοιτάζει και ο πρόεδρος της Επιτροπής, όχι γιατί περιμένει απάντηση, αλλά χαμογελάει με νόημα. Ο πραγματισμός, ο ρεαλισμός είναι το βασικό ζήτημα εδώ δεν μπορούμε να επιβάλλουμε λύσεις σε κράτη-μέλη. Ε, είδατε τις ε, αντιδράσεις των κρατών μελών. Ο κύριος Σούλικ από την ομάδα μας έθεσε ένα πολύ σωστό ερώτημα. Το ερώτησε τι κάνουν οι πολιτικοί όταν ε, η πλειοψηφία σε ένα κράτος μέλος δεν θέλουν μια λύση που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κύριος Πιτέλα τι είπε. Είπε ο κύριος Πιτέλα ότι πρέπει να δεχθούν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φοβούμαι ότι δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Ο σωστός τρόπος είναι όλα τα κράτη-μέλη μαζί να αποφασίσουν τι θέλουν όλα μαζί να κάνουν. Γιατί όλα τα κράτη-μέλη θέλουν λύσεις και όχι λύσεις που τους έχουν επιβληθεί. Και τώρα για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Φερχόστατ. Συνάδελφοι, υπάρχει ένα ρητό που λέει όταν παίζεις με τη φωτιά, μπορείς να περιμένεις και να καείς. Πρέπει να σας πω, εγώ αυτή την εντύπωση έχω ότι ακριβώ αυτό συμβαίνει με τη συμφωνία με την Τουρκία. Γιατί προσπαθήσαμε να, να λύσουμε ένα σωρό προβλήματα με τον ηγέτη της Τουρκίας, τον κύριο Ντογάν και τι έκανε πριν δύο μέρες. Έδωσε οδηγίε στην γερμανική κυβέρνηση να ασκήσει διώξει κατά ενό παρουσιαστή στην τηλεόραση, τον κύριο Μπένερμαν, για, την σατυρά... για τη σάτυρά του εναντίον του προσώπου του. Αυτό που έχει κάνει ο κ. Μπέρνεμαν δεν είναι ούτε για το δικό μου χιούμορ πολύ ευχάριστο, αλλά ζούμε σε ελεύθερη κοινωνία. Πρέπει να είναι ελεύθερη άσκηση κριτική και η σάτυρα. Πληρώνουμε για την ελευθερία μα και είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να πληρώσουμε για αυτήν. Για να επανέλθω λοιπόν στον κύριο Ερντογάν, ήδη το έχουμε δώσει τα κλειδιά για τις πύλες της Ευρώπης. Και τώρα τι θα κάνουμε. Θα του ε, εγχειρήσουμε και τα κλειδιά για τα στούντιο, τα τηλεοπτικά, για να αναλάβει και τα μέσα μαζικής μας ενημέρωσης. Δεν μου κάνει εντύπωση που συμβαίνει αυτό. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Εάν ε, βρεθείτε στη θέση να αφαιθείτε στο έλεος κάποιου, όπως του κυρίου Ερντογάν, και αναθέσετε εξωτερικώς, ε, διώξτε τι ευθύνε σα γιατί στείλετε σε μια χώρα όπως η Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, τι να σα πω, αυτό είναι μόνον η αρχή αυτού που θα ονόμαζα ε, πολιτική τουρκοπάζαρου. αυτό που έχει πει ο κύριος Ερντογάν στην Τουρκική Βουλή είναι ότι θα ακυρώσει την συμφωνία θα την αναστείλει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν μέσα σε δύο μήνες δεν απελευθερωθεί το καθεστώς των θεωρήσεων που ζήτησε. Ε, και ασχέτω αν θα τηρήσει τη δική του πλευρά τη συμφωνία ε, και ε, αν, πρέπει να δούμε αν θα συμμορφωθεί με τι ειδικέ μα συνθήκε για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Άρα εμεί έχουμε φέρει το σε αυτού μα να, εκτιθέμεθα στον κύριο Ερντογάν και να είμαστε ανυπεράσπιστοι στα χέρια του. Έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει το ίδιο με τον Πούτιν που χρησιμοποίησε την ενέργεια. Ο ε, Ερντογάν τι χρησιμοποίησε τους φτωχούς μετανάστες. Αυτό συμβαίνει. Και δεν το λέω αυτό ελαφρά την καρδία πρέπει να σας πω. Η πρώτη απόδειξη είναι ότι η Τουρκία ε, που ήταν μέρος της συμφωνίας κύριε Γιούνκερ ε, δεν τηρεί τη συμφωνία. Οι ίδιοι Τούρκοι δεν την τηρούν. Στην Τουρκία πρέπει να αλλάξουν την νομοθεσία τους πρέπει να άρουν τις εδαφικές τους ε, απαιτήσει βάσει των, ε, της συνθήκης της Γενέβης και θα πρέπει οι πρόσφυγες να έχουν άσυλο στην Τουρκία. Δεν τους το δίνουν και αρνούνται και να το κάνουν. Επιπλέον και ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι εκθέσεις μας, τα στοιχεία μας, κανείς δεν τα αναφέρει, συζητάμε εδώ πέρα και έχουμε στοιχεία από την Διεθνή Αμνηστία που λένε ότι η Τουρκία στέλνει τους μετανάστες πίσω, τους πρόσφυγες πίσω στην Συρία ενάντια στο διεθνές δίκαιο και χθε ε, επιβεβαιώθηκε από το Ολλανδικό τηλεοπτικό κρατικό κανάλι σε σχετικό πρόγραμμα ότι οι τουρκικές αρχές το κάνουν αυτό επισήμως. Η ερώτησή μου προς εσάς κύριε Τούσκ είναι γιατί δεν το εξετάζετε το θέμα αυτό, γιατί δεν το ερευνάτε, αληθεύει. Και αν ευσταθεί, μπορούμε να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια συμφωνία που αντίκειται στην ε, διεθνή νομοθεσία και στο διεθνέ δίκαιο και στι δικέ μα υποχρεώσει. Τι κάνετε, τι έχετε να μου απαντήσετε, πώ ε, κάνετε έρευνα για το θέμα αυτό. Αληθεύουν αυτά που είπε η Διεθνή Αμνηστία και το κρατικό κανάλι τη Ολλανδία χθε. Και τρίτο στοιχείο. Α μην αυταπατώμεθα αληθεύει ότι η συμφωνία ε, είναι αυτή που είπατε για τα ελληνικά σύνορα. Δεν είναι 700 την ημέρα αυτοί που έρχονται, είναι 50. Χθε όμως η, το Ιταλικό προξενείο ε, διέσωσε όχι 50 ανθρώπους αλλά 2.504 ανθρώπους Ποιο είναι το αποτέλεσμα λοιπόν αυτή τη διάσωση από την ακτοφυλακή. Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για τη συμφωνία, μπορούμε να αναφέρουμε αριθμούς, αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά από τους 50 στους 250 ε, και στους 1000, ε, 2154. Αυτή είναι η θέση μας, αυτή είναι η ελευθερία μας που την αφήνουμε έτσι στα χέρια του Ερντογάν. Αυτό θέλω να πω, ότι αντί να συζητάμε εδώ για μια συμφωνία που κατά την άποψή μου δεν λειτουργεί, θα πρέπει λιγάκι να συμμαζευτούμε εδώ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας εδώ. Και αυτό κατά την άποψή μου σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά ζήτησε αριθμό ανδρών από τα κράτη-μέλη. 400 ζητήσαμε και μόνο 37 ε, στάλτηκαν στην Ευρώπη. 472 ε, αξιωματούχοι για την ε, μετανάστευση ζητήθηκαν και τελικά απεστάλησαν μόνο 31 προς την Ελλάδα και την Τουρκία, κύριε Τούσκ. 500 αξιωματικούς ζητήθηκαν, ζήτησαν από την Ελλάδα και την Τουρκία και στείλαν μόνο 330. 2.500 ουσιαστικά έχουν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πόσο στείλαν τα κράτη-μέλη. 400 λίγο πολύ, κύριε Τούσκ. Τόσοι διατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η συμφωνία που πετυχαίνει. Εγώ τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Χρειαζόμαστε απελπισμένα την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και πρέπει να συμφωνήσουμε ώστε να λειτουργήσει. Και απελπισμένα πρέπει να λειτουργήσει και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, όπως και ο κύριος Πιτέλα, στηρίζω από την ομάδα μου την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να υλοποιηθεί στο δυνατόν γρηγορότερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τους λαθρέμπορους, ένας τρόπος υπάρχει να επιτρέψουμε να επανέλθει η νόμιμη μετανάστευση στην Ευρώπη. Είναι ο μόνο τρόπο να αντιμετωπίσουμε του διακινητέ, είτε στην Τουρκία είτε στη Βόρεια Αφρική. Ευχαριστώ. Κύριε Φερχόφστατ, ο κύριος Κάβα θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Το δέχεστε? Ευχαριστώ κύριε Φερχόφστατ. Μπορεί να διαφωνούμε πολιτικά, αλλά συμφωνώ μαζί σας, ε, συμφωνώ γιατί αυτά που λέτε είναι σωστά. Είπατε αυτό που είχε πει ο Ρόι Τζένκινς, ε, πρώην Βρετανός πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να έχουμε μια συνεπή στάση έναντι της Βρετανικής ε, θέσης στην Ένωση. Είστε εντελώς εντός ή εντελώς εκτός. Συμφωνείτε λοιπόν ότι τα μηνύματα από το σώμα μας μοιάζει να είναι ότι τελικά έχει λήξει η υπομονή, έχει τελειώσει η υπομονή των Βρετανών πολιτών με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Κύριο Φερχόφστατ, χαίρομαι για το βρετανικό σας χιούμορ, αλλά θεωρώ ότι είναι περισσότερο για τον κύριο Καμάλ που είναι ειδικό για αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για την ε, ενιαία Ευρωπαϊκή Αριστερά, η κυρία Τσίμα. Κυρίες και κύριοι, Κύριε Πρόεδρε, όσοι ε, μιλήσατε προηγουμένως για το σύστημα, νομίζω πως δεν λειτουργεί το σύστημα. Νομίζω ότι η κοινή γνώμη κάνει πολύ σκληρή κριτική. Για τη συμφωνία με την Τουρκία, εσείς λέτε ότι ναι, έχουμε κάποιες αμφιβολίες για την ηθική και νομική βάση, αλλά από την άλλη πλευρά λέτε ότι αυτά καταφέραμε, αυτό μπορούσαμε να επιτύχουμε. Και δεν υπάρχει καμία πανάκια, μα δεν λειτουργεί το σύστημά σας. Πρέπει να κάνετε πολύ περισσότερα. Δεν μπορείτε να πείτε δεν θα έχουμε ποτέ την καλύτερη λύση ε, και μπορεί να μην πηγαίνει τόσο καλά, δεν είναι τόσο θαυμάσια και από την άλλη μεριά να αποσιωπάτε την πραγματική κατάσταση. Ο κύριος Βέιμπερ έχει αυτές τις, ε, αυτούς τους εμφιάλτες ε, και βλέπει μπροστά του το φάντασμα του κομμουνισμού, του Τσίπρα ή άλλων πρέπει να πω ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν πια ποια είναι η πραγματικότητα. Εμείς ως Ένωσης, εμείς καταστρέφουμε την Ελλάδα με κάθε απόφαση για μεταφορά, για επιστροφή ε, μεταναστών στην Τουρκία θεωρούμε ότι είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία. Ενώ επί λέγαμε στην Ελλάδα ότι δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τα, τα εξωτερικά σύνορα, δεν καταλάβατε πόσο μακριά είστε από την πραγματικότητα στη χώρα. Ο κ. Φερχόφστατ μας διηγήθηκε τι σημαίνει η εφαρμογή τη συμφωνία και τι συγκεκριμένη βοήθεια πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έχουν υποσχεθεί και τι έχει δοθεί. Επιβάλλουμε μια διαδικασία καταγραφής των αιτήσεων στην Ελλάδα η οποία είναι σε ελάχιστες προδιαγραφές. Πρόκειται για μείωση των προδιαγραφών για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Και αν αυτό θα πρέπει να είναι το επίπεδο εξέτασης ε, στο μέλλον και αν αυτό θα είναι το πρότυπο για περαιτέρω συμφωνίες, τότε μπορώ να σας πω ότι απομακρυνόμαστε από τις αρχές μας, από τις απαιτήσει μας για ανθρωπιά και αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να είναι σαφές και να υποθεί σαφώς. Ένα είναι να υπάρχουν ανεπάρκειες, αλλά είναι άλλο να κάνουμε σαν να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση και ότι οποιοδήποτε επικρίνει είναι κακόβουλος. Και πρέπει να σας πω ότι Είμαστε κατά του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται τώρα την Τουρκία. Την Τουρκία του Ερντογάν και τη θεωρείται ασφαλή τρίτη χώρα. Ακόμη και η επιστημονική υπηρεσία του Γερμανικού Κοινοβουλίου εξέφρασε αμφιβολίες. Για να είναι ασφαλής ε, μια τρίτη χώρα πρέπει να τηρούνται τα δικαιώματα των προσφύγων. Στην πράξη αυτό δεν γίνεται. Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία από τα μέση Ιανουαρίου έχουν επιστραφεί στη Συρία. Δεν έχουν κλείσει τα σύνορα. Μάλλον έχουν κλείσει τα σύνορα. Πυροβολούν τους πρόσφυγες. Και ότι έχουν ε, δολοφονηθεί και παιδιά. Πότε τα συζητάμε αυτά εδώ. Αυτό είναι το ερώτημα. Και το μόνο που μπορώ να σας πω είναι παρακαλώ να δημιουργήσετε μια ανοιχτή πολιτική ασύλου και να τονίσετε και τις ευθύνες των κρατών μελών πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Για τους πράσινους, η κυρία Χάρμς. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η τελευταία συμφωνία κορυφής είναι ότι από κοινού θα εργαστούμε για να υπάρξει ε, σωστή κατάσταση και κράτος δικαίου και τήρηση των κανόνων για την ε, εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Θέλουμε επίσης να υπάρχει αξιοπρέπεια για αυτούς που ζητούν άσυλο. Αλλά αυτό που συμβαίνει εδώ και εβδομάδες και που το διαπιστώνουμε κάθε μέρα και το ακούμε κάθε πρωί και κάθε βράδυ στις ε, ειδήσει. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα λοιπόν. Αυτό δείχνει ότι ναι υπάρχει κάποια τάξη αλλά ανθρωπιά και δίκαιο καθόλου. Για παράδειγμα είδαμε στην Ιδωμένη αυτά που μας είπε ο Νόρμπερτ Μπλουμ, πρώην υπουργό Γερμανός, ο οποίος ρώτησε πάντα πότε επιτέλους θα εφαρμόσετε τις αρχές της ανθρωπιάς, πότε θα εφαρμόσετε τους νόμους και Του είπαν κύριε Τουις που λέτε πως δεν είναι 100% αυτά που του είπαν είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε καθόλου για εφαρμογή των κανόνων και κράτος δικαίου στις διαδικασίες. Και αυτό είναι η κύρια ευρωπαϊκή μας ευθύνη πριν αναφερθούμε στις δυσκολίες που υπάρχουν στην Τουρκία. Πρέπει εμείς εδώ στην επικράτειά μας, στο σπίτι μας, στην Ένωση να είμαστε σε θέση να παράσχουμε κράτος δικαίου για τους πρόσφυγες. Αν μπορούν να γίνουν πριν δημιουργήσουμε την συνοριοφυλακή και την ακτοφυλακή, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, αν μπορεί να γίνει 100% δεν είμαι σίγουρη, αλλά η σημερινή κατάσταση να συνεχίσουμε να τη δεχόμεθα δεν είναι δυνατόν. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνοηθεί με τις ελληνικές αρχές και τους Έλληνες πολιτικούς να αλλάξουν την κατάσταση. Γιατί για μένα αυτά που συμβαίνουν τώρα συνολικά δυσφημούν τη συνολική πολιτική ασύλου και δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές για να εκφοβήσουμε αυτούς που θα ήθελαν να έρθουν στην Ευρώπη. Τώρα στην Τουρκία, εφόσον υπάρχει αυτή η συμφωνία για τους πρόσφυγες, έχουμε και εμείς αναλάβει λοιπόν ευθύνη για το τι συνθήκες επικρατούν στην Τουρκία το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και εβδομάδες εφόσον λάβαμε τις πληροφορίες ότι στέλνονται πίσω στη Συρία πρόσφυγες θα έπρεπε λοιπόν από τότε που το μάθαμε να έχει διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν ισχύει και αν ισχύει τότε θα έπρεπε να επανεξετάσουμε τη συμφωνία και ενδεχομένως να την αναστείλουμε. Και τώρα να απευθυνθώ στον συνάδελφο Φερχόφστατ. Για τα θέματα της ε, ακτοφυλακής και της σύνοροφυλακής συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υποκλεινόμεθα μπροστά στον πρόεδρο Ερντοάν. Όπως μου είπαν και διάφοροι της αντιπολίτευσης και στο Κουρδιστάν και στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, πιστεύω λοιπόν ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί τις απαιτήσει μας για κράτος δικαίου στην Τουρκία και έχει κατακτήσει το δικαίωμα να θέλει να βελτιωθεί η κατάστασή της. Δεν πρέπει λοιπόν να δυσφημίσουμε τις προσπάθειες που κάνει. Γιατί αν δούμε συνολικά την κατάσταση στην Εγγύη και Μέση Ανατολή και αν δούμε ε, απλά και μόνο τη γεωγραφική θέση της Τουρκίας και την κοινή μας ιστορία, δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να τους δυσφημίσουμε. Και τώρα, η ελευθερία του λόγου και της τέχνης δεν ε, θα αποφασιστεί από τον Ερντοάν στη Γερμανία. Νομίζω ότι η χώρα μου είναι αρκετά δυνατή για να μπορέσει να τηρήσει τις αρχές της αυτήν την αντιπαράθεση με τον Ερντοάν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για το EFDD τώρα, ο κύριος Φάροντς. Ευχαριστώ. Εκπλήσωμαι που βρισκόμαστε εδώ στον οίκο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και αυτό το πρωί θα έπρεπε να γιορτάζουμε για το Ολλανδικό δημοψήφισμα την περασμένη εβδομάδα που είπαν όχι στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Ολλανδοί, όχι στη συμφωνία με την Ουκρανία. Και αν ήταν ε, θέμα και η συμφωνία με την Τουρκία, θα είχαν πει όχι στην προσχώρηση τη Τουρκία. Ήταν νίκη τη δημοκρατία αυτό λοιπόν. Αλλά όλο ιδιαίτερο ήταν νίκη για την Kingpile, ένα, μια ομάδα νέων που κατάφεραν να συγκεντρώσουν 120.000 υπογραφές υπέρ της άμεσης δημοκρατίας. Έτσι θυμόμαστε τον, ε, τον κύριο Τζαστελόντιο που ήταν ο ιδρυτής του κινήματος των Πέντε Αστέρων στην Ιταλία ε, Βεβαίω, εντωμεταξύ, μα είπε ο κύριο Γιούνκερ ότι αν είχαν ψηφίσει όχι οι Ολλανδοί θα ήταν καταστροφή. Σήμερα το πέρασε στο. δεν το ανέφερε καθόλου. Και ο κ. Φαντόρομποϊ, ο φίλο μου, ο προκατοχός σα, έλεγε ότι πρέπει να προχωρήσουμε ε, ακόμη και αν οι Ολλανδοί έχουν κάποιε αντιρρήσει. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε. μεγάλε δυνάμει κάνουν ό,τι μπορούν για να αγνοήσουν τη βούληση των Ολλανδών, του Ολλανδικού λαού μας. Τα πράγματα αλλάζουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτά τα θεσμικά όργανα μπορούν να επιβιώσουν ε, στην τεχνολογία του 21ου αιώνα. Νομίζω ότι η βούληση των πολιτών αλλάζει την πολιτική και τα πολιτικά πράγματα με τρόπο που θα σα κάνει όλου εδώ πραγματικά να φοβάστε και έτσι θα έπρεπε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το δικό μα δημοψήφισμα. Και όλα τα μάτια είναι στραμμένα προ τη συμφωνία με την Τουρκία. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν τώρα να συμβαίνει είναι τα αφεντικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, κάνουν αδέξιες χειρονομίες μπροστά στον κύριο Ερντογάν ε, με, καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα και βλέπουμε τον κύριο Γιούγκερ να μας λέει σήμερα το πρωί ότι Έχουμε μια καλή συμφωνία. 1,8 εκατομμύρια έχουν έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση του τελευταίου 18 μήνε και εμεί λέμε ότι 300 επανακαταστήσαμε. Δεν θα έλεγα το σύστημά σα λειτουργεί και πολύ καλά. Η μόνη ομάδα που θα ε, ικανοποιηθεί με όλα αυτά είναι η ISIS έχουν ε, καταφέρει 5.000 από τους μαχητές τους να τους φέρουν στο ευρωπαϊκό έδαφος βάσει των στοιχείων της Europol. Αυτό θα έπρεπε να ε, κάνει τις ραχοκουκαλιές μας να αναρριγούν. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι στο δημοψήφισμα της Μεγάλης Βρετανίας θα πρέπει να δείτε τι θα γίνει γιατί θα ψηφίσουμε για το Brexit και θα θέλουμε να γίνει και γοργά. Αυτό ε, έγινε και στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα. Μάχη του λαού κατά των πιλωτικών. Εσεί μπορεί να έχετε στα χέρια σα τα πολλά τα λεφτά και τι μεγάλε εταιρείε. Εμεί όμω έχουμε ένα στρατό από blogger μαζί μα. Και η βούληση των πολιτών θα υπερισχύσει. Αυτό το μέρο δεν θα επιβιώσει. Ο κύριος Έριξον θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Φαράζ που κάθεται πίσω από τη Βρετανική σημαία. Δεν νομίζετε ότι για πολλούς Βρετανούς αποτελεί ντροπή κάποιος που μιλά καθήμενος πίσω από μια Βρετανική σημαία, μιλά υπέρ ε, ενός δημοψηφίσματος όπου ο μόνος νικητής θα είναι ο κύριος Πούτιν ο οποίος επιχαίρει γιατί η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη τώρα για τη συνεργασία με την Ουκρανία ο κ. Φαράζ. Δεν είμαι υπέρμοστο του κ. Πούτιν, αλλά ούτε και υπέρ του πολέμου με τον κύριο Πούτιν. Νομίζω θα ήταν μια ανόητη ιδέα ενθαρρύνουμε την κατάρρευση ενός διαφθαρμένου ηγέτη που όμως είχε εκλεγεί δημοκρατικά στην ε, Ουκρανία νομίζοντας ότι ε, αν χτυπήσουμε την ρωσική αρκούδα δεν θα αντιδράσει καθόλου. Πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τις εθνικές μας δημοκρατίες. Κύριε Έριξον, θέλουμε να συνεργαστούμε, να έχουμε εμπόριο με τους γείτονές μας, να είμαστε φίλοι, αλλά αυτό που δεν θέλουμε είναι αυτή η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης και τον Εθνικό Ύμνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να είμαστε φίλοι γείτονες. Äh, e Ο κ. Βιλίμσκι για την ομάδα των Εθνών και της Ελευθερίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έχοντας ακούσει τους προηγούμενους ομιλητές από τα προηγούμενα κόμματα και τον κύριο Πιτέλα ασκώντας ε, κριτική ε, στην Αυστρία που πήρε μόνο 36 μετανάστες θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ε, ήρθαν 90.000 πέρυσι και με την ε, βοήθεια του ε, καγκελάριου ε, Φάιμαν κατάφεραν οι διακινητές να αφήσουν ένα εκατομμύριο να περάσει στη Γερμανία μέσω της Αυστρίας. Γι' αυτό διαφωνώ με τα επιχειρήματά σα και για τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο επίση θέλω να πω δύο λόγια γιατί ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κύριο Μάνφερ Βέμπερ ε, τα λόγια ε, του βαβαρού πρωθυπουργού. Ευτυχώ που στην Γερμανία υπάρχει το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία που σιγά σιγά καταλαμβάνει τους ψηφοφόρους και της δικής σας πολιτικής ομάδας και για αυτά που είπαν οι πράσινοι επίσης θέλω να πω ότι θέλουμε να έχουμε δημοκρατικές ε, αποφάσεις στην Ευρώπη αλλά τι κόμμα είστε εσείς, είστε ένα κόμμα ε, ε, που ξεκίνησε από τη βάση αλλά θέλετε να μην αφήσετε το λαό να αποφασίζει για τα δημοκρατικά του δικαιώματα. Αυτή η συμφωνία με την Τουρκία κινείται προς εντελώς λάθος κατεύθυνση και είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά και να μην βλέπουμε τι συμβαίνει στην Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τους Κούρδους, για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Δείτε ε, τι ζητεί ο λαός. Στην Ολλανδία λήφθη μια σωστή απόφαση κατά της ασφαλμένης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το σωστό μοντέλο για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάλτσο ευχαριστώ πρόεδρε. η συμφωνία μεταξύ ευρωπαϊκής ένωσης και τουρκίας ορίζει ότι μπορούν νόμιμοι μετανάστες να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στις Ευρωπαϊκές Ένωσης λοιπόν φαίνεται να χωρίζουν τους μετανάστες σε καλούς και κακούς. Όμως αυτοί που φτάνουν με ένα φεριμπότ στην Ελλάδα χωρίς έγγραφα αποφασίστηκε ότι πρέπει να στέλνονται πίσω. Όταν όμως υπάρχει ένα σοβαρό, ένας αριθμός ε, ανθρώπων που του στέλνει με τα χαρτιά του η Τουρκία στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι είναι καλοί μετανάστε. Τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκέ κοινωνίε λοιπόν, Θα χτίσουμε παράλληλε κοινωνίε που θα μπορούν αυτοί οι μετανάστε να ενταχθούν κανονικά και θα αποκλείσουμε από αυτέ του μετα... τρομοκράτε. Δεν μπορώ να δω πώς αυτά μπορούν να υλοποιηθούν. Πρέπει να κοιτάξουμε τι θα γίνει με τους μετανάστες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να λέμε στην Αυστραλία και στον Καναδά τι θα κάνουν. Και το είπε και η κυρία Τσίμερ εδώ πέρα, μόλι τώρα. δεν είμαστε απλώς μια Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Έχουμε τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να αποφασίζει και το μεγαλύτερο μέρος αυτού δεν θέλει τους μετανάστες στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρόιλ. Κύριε Πρόεδρε, Δεν καταλαβαίνω πλέον τον κόσμο. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και έχουμε εκνευριστεί ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένα μέτρα για τους πρόσφυγες. Η κύρια δουλειά μας είναι να ε, βοηθήσουμε τους πρόσφυγες και στραφήκαμε κατά του Συμβουλίου και είπαμε αυτοί οι ανόητοι, αυτοί οι εγωιστές δεν αποφασίζουν. Αποφασίστε. Και αντί γι' αυτό η κυρία Τσίμερ τώρα που λύθηκε μια απόφαση και θα μπορούσαν να πούν ότι επιτέλους έγινε κάτι, απλώς γκρινιάζουν. Αυτό κάνουμε. Γκρινιάζουμε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη. Η σημαντικότερη φράση που ακούστηκε σήμερα το πρωί ήταν η πρόταση του κυρίου Τίσκ αναλάβαμε την ευθύνη μας. Τα κράτη-μέλη ανέλαβαν την ευθύνη τους και είπαν θα κάνουμε κάτι. Φυσικά δεν είναι τέλεια λύση. Δεν ισχυριζόμεθα κάτι τέτοιο. Βεβαίως ε, πολιτική αυτό σημαίνει. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν τέλειες λύσεις. Υπάρχουν μόνο βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, είναι μια δυνατότητα, είναι συγκεκριμένη βοήθεια. Έχουμε και η δυνατότητα επιστροφής ορισμένων. Ορισμένοι λένε ότι έχουμε παραδοθεί στην Τουρκία, μα αυτά είναι ανοησίες. Αντίθετα, με αυτές τις επικρίσεις εγώ από την αρχή Ήμουν και είμαι κατά τη ένταξη τη Τουρκία. Ορισμένοι άλλαξαν γνώμη και λένε βεβαίω. Βεβαίω αύριο να ενταχθούν. Ο ένα λέει ότι είναι θαυμάσια η Τουρκία και μετά λέει όταν δεν συμφωνεί με κάτι που έκανε ότι είναι απέσια. Αυτά που είπε η κυρία Χάρμς ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Να πει ότι πολλά δεν ε, με βρίσκουν ε, ε, σύμφωνοι. Και εγώ συμφωνώ και εμένα πολλά δεν με βρίσκουν σύμφωνα από αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Αλλά ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είπε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την Τουρκία. Και τώρα υπάρχει. Αυτό είναι ένα βήμα. Θαυμάσιο. Θαυμάσιο. Κάναμε ένα βήμα το επόμενο. Αλλά να προσέξουμε να μην κάνουμε και άλλα λάθη. Βεβαίω. Αλλά να κάνουμε τέτοιε επικρίσει. Το Κοινοβούλιο, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα είναι πλέον αξιοπρεπή θεσμικό οργανισμό. Αν γκρινιάζουμε και είμαστε κατά πάντων. Πρέπει να βοηθήσουμε συγκεκριμένα τους ανθρώπους. Γι' αυτό μας πληρώνουν, γι' αυτό μας έστειλαν εδώ. Έχει ζητηθεί μπλε κάρτα για σας κύριε Ρόιλ από τον κύριο Λάμσδορφ. Τη δέχεστε? Ο κύριος Λάμσδορφ. Αγαπητέ Χέρμπερτ. Ας πούμε ότι είναι καλή η συμφωνία. Και εγώ την επικρίνω βεβαίως αλλά όντω είναι βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση, τότε πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του στα κράτη-μέλη. Το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα είπε στην Ελλάδα, Ιωνία, υπάρχουν δύο ή τρει υπηρεσία ασύλου τη Γερμανία και οχτώ ακόμη θα πάνε. 30 Γερμανία αστυνομική. Συμφωνεί ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε τη. Ότι αυτή η συμφωνία, εφόσον στηρίζεται υπεύθυνα πρέπει να στηριχθεί και με επαρκές προσωπικό και ότι αφήνουμε συγκεκριμένα η Μέρκελ και ο Ντεμεζιέρ τον Τουίσκ και τον Γιούγκερ να λύσουν όλα τα προβλήματα. Ρόιλ, ναι. Βεβαίω και εγώ θα ήθελα να βοηθήσουν περισσότερο και να στείλουν περισσότερο προσωπικό όπω έχουν δεσμευτεί. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δυστυχώ δεν είναι τόσο απλό ορισμένε φορέ. Όποιο έχει εργαστεί σε διοίκηση το ξέρει. Φυσικά αυτά τα οποία υποσχόμεθα πρέπει να τα τηρούμε. Βεβαίω για όλα τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη επίσης πρέπει να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους που έχουν πει ότι θα δεχθούν πρόσφυγες. Όλα σωστά. Όλα σωστά. Το προσωπικό που έχουμε υποσχεθεί πρέπει να το στείλουμε. Σαφές. Η κυρία Φαγιόν. Danes imamo sporazum s θα ήθελα να μπορούσα σήμερα να πω ότι έχουμε μια καλή συμφωνία με την Τουρκία, μια συμφωνία που λειτουργεί και που έχει σωστή νομική βάση. Δυστυχώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Και ε, όλο και περισσότερο έχω την εντύπωση ότι δεν είναι καλή συμβαστική λύση. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω άλλη εναλλακτική λύση. Θα ήθελα να λειτουργεί η συμφωνία με τρόπο ώστε να γίνονται σεβαστά τα βασικά δικαιώματα των προσφύγων και ε, θέλουμε να αποφύγουμε να συνεχίζεται η κατάσταση με τους διακινητές που φέρνουν ε, συνέχεια μετανάστες στα ελληνικά σύνορα και ε, αυτό που ακούμε ότι από την Τουρκία επιστρέφονται πρόσφυγες στην Συρία. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, βλέπουμε πόσο κακή είναι η κατάσταση με τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Τουρκία. Ξέρουμε πόσο μας σοκάρουν οι εικόνες από τα hot spots στην Ελλάδα που έχουν μετατραπεί σε κλειστά στρατόπεδα κράτησης. Θα θέλαμε να έχουμε ε, μια σωστή συμφωνία με την Τουρκία που να εγγυάται το κράτος ε, δικαίου. Ε, Εάν ε, δεν ε, λειτουργήσουν τα προγράμματα επανεγκατάστασης, ε, εμείς φέρουμε την ευθύνη, γιατί θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να μην χτίζουμε φράχτες στα σύνορα, να σταματήσουμε το εμπόριο ανθρώπων, τον εμπόριο ανθρώπων γυναικών και παιδιών, και έχουμε τώρα μια φιλόδοξη προσπάθεια να μεταρρυθμίσουμε τον κανονισμό του Δουβλίνου και ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε. Ο κύριος Έτεριτς θέλει να κάνει μια ερώτηση. Καλημέρα. Ευχαριστώ που δέχεστε την ερώτησή μου. Θα μπορούσατε να διευκρινίσετε ή μαζί με τον επικεφαλή σας, τον κύριο Πιτέλη, να συμφωνήσετε στα σχόλια που έκανε προηγουμένως. Συμφωνείτε μαζί του ότι είναι εγωιστικό εκ μέρους των κρατών μελών να αποφασίζουν πόσους πρόσφυγες θα δεχθούν. Συμφωνείτε μαζί του ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δέχονται κάποιου, κάποιους αριθμούς προσφύγων και να τους επιβάλλεται κάτι τέτοιο. Και ε, η έλλειψη ε, σεβασμού ε, προς άλλους ηγέτες ευρωπαϊκών κομμάτων πιστεύετε ότι είναι αποδεκτό. Ε, Αγαπητέ συνάδελφε, με αυτό που συμφωνώ είναι ότι σήμερα αυτό που θέλουμε είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν, συμφωνεί και λειτουργεί. Και συμφωνώ με όλου οι οποίοι λένε ότι πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τι ευθύνε του για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα κατανομή των προσφύγων. Μπορεί να μην λειτουργεί το σύστημα μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση γιατί πολλά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλαμβάνουν τι ευθύνε του. Και όταν δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι είναι περιτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και σας παρακαλώ όλους να αναλάβετε τις ηθικές σας ευθύνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τον Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξαναγκάστηκε από τα γεγονότα να ε, ε, λάβει τις αποφάσεις του, αλλά ήδη είχαμε και άλλες εξέλιξεις στις τρομακτικές επιθέσεις της Βρυξέλλας στις 22 Μαρτίου και τα αποτελέσματα του Ολλανδικού Δημοψηφίσματος. Στην πρώτη περίπτωση, Πρόεδρε, ε, ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο τι θα, μέτρα θα λάβει για να εξασφαλίσει ότι είναι ασφαλής τα θεσμικά, ασφαλή τα θεσμικά όργανα όπου, για τα οποία είναι υπεύθυνο, καθώ και το προσωπικό που εργάζεται εκεί και οι επισκεπτόμενοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ω προ τη διοικητική δουλειά των θεσμικών οργάνων. Και δεύτερον, το δημοψήφισμα στι κάτω είναι πρόβλημα για την κοινή πολιτική ασφάλειας και την κοινή εξωτερική πολιτική. Χρειάζονται εδώ κάποιες νέες ιδέες για το πώς θα χειριστούμε πλέον την Ρωσία. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για συνεργασία με την Ρωσία, ούτε μπορούμε να κοιτάμε μόνο προς τον Νότο. Και ένα ακόμα στοιχείο η ε, ε, βίαιη παρέμβαση στις πολωνικές υποθέσεις και το ψήφισμα που θα εγκριθεί σήμερα με το πονίδι στο περιεχόμενό του νομίζω ότι ουσιαστικά ε, παραπλανεί τον κόσμο. Κυρία Γιάκον Σάρη, μπορείτε να απαντήσετε σε ερώτηση σε κάρτα. Ευχαριστώ. δεν κατάλαβα καλά την σχέση μεταξύ Ολλανδικού Δημοψηφίσματος, Ρωσίας και Πολωνίας. Μιλάμε για πολύ σοβαρά ζητήματα εδώ. συζητούμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα τη ε, τεράστια ροής μεταναστών και των ασύλου και πώς θα διασφαλίσουμε δίκαιη μεταχείριση. Δεν πρέπει να συγκεντρωθείτε στο θέμα που συζητιέται Νομίζω ότι αυτό πραγματικά είναι το πλέον ε, μεγάλο πρόβλημα για όλους στην Ευρώπη. Κυρία μου, δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς ε, σας δόθηκε μέσω της διερμηνίας η παρέμβασή μου μέσα από τις διάφορες γλώσσες. Ωστόσο, πιστεύω ότι το μέλλον θα μας δείξει. Θα δείξει ότι υπάρχει σαφής διασύνδεση μεταξύ όλων αυτών των ζητημάτων. Αναφερόμουν επίσης στα διοικητικά, τις διοικητικές δυνατότητες να επιλύσουμε προβλήματα μετά τις δημοκρατικές επιθέσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Λάμπστορφ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, Πιστεύω ότι ένα βλέμμα στο χάρτη δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία παίζει ένα κεντρικό ρόλο, έχει τρία εκατομμύρια πρόσφυγες. Αυτό το δείχνει μια πρώτη ματιά στο χάρτη. Ε, μια δεύτερη ματιά στο χάρτη δείχνει ότι υπάρχει η οδός της Μεσογείου και ο κύριος Καμάλ έχει δίκιο που λέει ότι το καλοκαίρι έρχεται με τις μεγάλες ροές προσφύγων. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει όμως είναι ότι η υλοποίηση ε, αυτής της συμφωνίας πρέπει να γίνει με τρόπο ανθρωπιστικό και δίκαιο. Δεν θα πρέπει να ε, εγκαταλείψουμε την ε, εξατομικευμένη εξέταση των δικαιωμάτων των προσφύγων. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ε, βοηθήσουμε ε, αυτές τις προσπάθειες στα, για τον έλεγχο στα σύνορα. Έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε περισσότερους υπαλλήλου για να αποφύγουμε τις τραγωδίες στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κυρία Βεργιά. Ευχαριστώ η Ευρώπη προτιμά να μετατοπίσει τους αστυνομικούς και παρά τους πρόσφυγες. Αυτό το είπε μια μη κυβερνητική οργάνωση της Ευρώπης και είναι η σύνοψη του τι έγινε στην ε, Ευρωπαϊκή Σύνοδο του Μαρτίου. Εδώ ε, στέλνουμε πίσω τους μετανάστες, ε, χωρίς κανέναν ελεγχό, ακόμη και σύρους, για προς που ξέρουμε ότι δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το γνωρίζετε Ευρωκοινοβούλιο, χωρίς καμία διεθνή προστασία. Άντρε, γυναίκες και παιδιά. Η υποδοχή μας και οι δυνατότητές έχουν φτάσει στο μηδέν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η ειδική μετανάστευση, λένε ότι δεν μπορούμε να ε, διακυβεύουμε την ε, ζωή των ανθρώπων αυτών και να του εκθέτουμε σε κάθε κίνδυνο. Εδώ ε, πρέπει μαζί με την υπατερμοστία και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις να συνεργαστούμε για να διασώσουμε ανθρώπινε ζωέ, να σεβαστούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αλλά αυτά μα προκαλούν όνειδος και ντροπή που είμαστε Ευρωπαίοι και υποτίθεται ότι περασπιζόμαστε αξίε όπω το άσυλο. Δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι ηθήνοντε να αντιμετωπίσουν την κοινή γνώμη. Δεν το δέχονται. Δεν αντιμετωπίζουμε όμω έτσι το λαϊκισμό. ρεαλιστέ είναι αυτοί που κοιτάζουν τον κόσμο είναι και ψάχνουν ε, λύσει χειροπιαστέ. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε ιδανικά. Ναι, θέλουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που δεν αφήνει του ανθρώπου να πεθαίνουν στη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η γεωγραφική ζώνη που οικονομικώ είναι η πλέον πλούσια. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε αλληλεγγύη και να φανούμε στο ύψο των προσδοκιών και τη ανθρωπιστική κρίση που διανύουμε αυτή την περίοδο. Ευχαριστούμε. Ο κύριο, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μιλάω από πλευρά της ομάδας ΙΦ που ανησυχεί πάρα πολύ για την ε, συμφωνία με την Τουρκία. Η συμφωνία αυτή δεν κάνει τίποτα για να λύσει την κρίση των προσφύγων. Αντί να δίνει μια κοινή ανθρωπιστική λύση, εγωιστικά τα κράτη-μέλη προσπαθούν απλώς ε, να κρύψουν από τους πολίτες της Ένωσης την κρίση και υποκρίνονται ότι η επιστροφή από την Τουρκία στη Συρία προσφύγων δεν έχει καμία σχέση με την Ένωση. Ξέρουμε τα δεινά και πόσο άσχημη είναι η κατάσταση στα τουρκοσυριακά σύνορα. Θα έπρεπε να έχουμε προτείνει μια φιλόδοξη και ενιαία προοπτική που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και την, ε, τον δίκαιο καταμερισμό ευθυνών. Επιπλέον η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα για τους πρόσφυγες. Δεν τους δίνει στοιχειώδεις συνθήκες καθεστώτος προσφύγων. Δεν είναι ασφαλής χώρα ούτε για τους πολίτες της η Τουρκία. Στην Τουρκία υπάρχει τρομερή καταπίεση και βία κατά των Κούρδων και άλλων μειονοτήτων. Η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει την λογοκρισία και να σεβαστεί την ελευθερία του λόγου και του τύπου. Η συμφωνία αυτή επιπλέον είναι παράνομη, γιατί διατυπώθηκε ως δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Προσπαθεί λοιπόν η Ένωση να αποφύγει τις υποχρεώσεις της με βάση το ενωσιακό δίκαιο συμπεριλαμβανομένης και της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων και παρακάμπτει και τις αρμοδιότητες του σώματός μας. Αρμοδιότητες συναπόφασης για θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να κάνει τα αναγκαία βήματα για να αποτιμήσει την ομιμότητα αυτής της συμφωνίας και όλων των αποφάσεων που απορρέουν και να την καταγγείλει στο δικαστήριο. Ευχαριστώ. Γαλάζια κάρτα από τον κύριο Φροντζουλίτσα. Τη δέχεστε. Θα απαντήσετε. Κύριε Τερικάμπρας. Κύριε Φροντζουλίτσα. Συνάδελφε, όπως υπόθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα αυτή, η συμφωνία με την Τουρκία δεν είναι τέλεια. Όμως φαίνεται σαν ένα βήμα πρόοδου. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι να κάνει εάν την ακυρώσει τη συμφωνία αυτή η Τουρκία. Είπε ο κ. Σοντοχάν την περασμένη εβδομάδα ότι αν δεν ε, πλέον τι υποχρεώσει τη ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να την καταγγείλει τη συμφωνία να πάσα στιγμή. Κοιτάξτε, συνάδελφε, τα πάντα φαίνεται ότι βρίσκονται στα χέρια τη Τουρκία πλέον, όλο το παιχνίδι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούμε εμεί να καταγγείλουμε τη συμφωνία. Η Τουρκία μπορεί. Αυτό τι δείχνει, ότι είναι παράνομη, παράξενη και ιδιόρυθμη η συμφωνία. Ευχαριστούμε κυρία Φαραρά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούσαμε σήμερα τον πρόεδρο τους και να μας λέει ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι τέλεια ότι κάναν ό,τι μπορούσαν για να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Συμβούλιο, ότι παραμένουν αμφιβολίε. Οι ίδιε αμφιβολίε ε, είναι αμφιβολίε που συμμερίστηκε και ο πρόεδρο Γιούνκερ. Όμω, εφόσον υπήρχαν αμφιβολίε, δεν χρειαζόταν να προχωρήσουμε. Δεν χρειαζόταν να προχωρήσουμε στην οδό των αμφιβολιών και των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρόκειται για αμφιβολίε που βασίζονται σε γεγονότα, στην ιστορία και σε πρόσφατα επεισόδια. Γνωρίζουμε βεβαίω ότι η λύση πρέπει να εξευρεθεί. Δεν ψάχνουμε το άγιο δισκοπότερο, ούτε την τελειότητα όπω μα είπε σήμερα ο πρόεδρο Τουρκ, Τουρκ συγγνώμη, αλλά θέλουμε μία λύση. Αυτό ε, που αναζητούμε είναι η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Στην ουσία όμω, ρεαλιστική αναθεώρηση, όχι αυτή που προτάθηκε πριν από λίγες μέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ε, έχει ίχνος ανθρωπιστικών διαδρόμων η λύση που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κι όμω θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη λαθρομετανάστευση υποτίθεται. Ε, λοιπόν, ας ψάξουμε μια νόμιμη εναλλακτική. Ας ψάξουμε μια νόμιμη εναλλακτική για να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Εάν αλλάξει ο κανονισμός του Δουβλίνου θα πρέπει να βασιστούμε και στην αρχή ότι η πρώτη χώρα άφηξη είναι αυτή που θα έχει τη μέγιστη ευθύνη για του ετούντε άσυλο. Εάν αλλάξει αυτή η αρχή θα αποφύγουμε μια χώρα να γίνει ένας τεράστιος καταβλισμό προσφύγων. Η Βαλκανική οδός έχει κλείσει. Στην Ιδωμένη η Μακεδονική αστυνομία έριξε ε, δακρυγόνα ε, προ τους μετανάστες κάθε παιδιά ε, μεταξύ άλλων και 2.000 είναι τα συνόδευτα ανήλικα που κατήγγειλε η Διεθνή Αμνηστία. Κατήγγειλε μάλιστα και την Τουρκία ως μη ασφαλή χώρα για τους πρόσφυγες. Η κατάσταση είναι καταστραφική. Ο συνολικός απολογισμός της συμφωνίας με την Τουρκία δίνει πολύ λίγα αποτελέσματα σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση των ανθρωπιστικών συνθήκων. Βεβαίω, αυτό που θα συμβεί δεν είναι ότι θα κλείσει η οδό των Βαλκανίων και δεν θα υπάρχει άλλη. Θα μετακινηθεί. Έρχονται μετανάστε από τη Μεσόγειο, στον Κρότονα. Έρχονται στο Ρέντο Καλάμπρια, στην Ιταλία. Ε, έχουμε λοιπόν απέναντί μας μια Ευρώπη με ελάχιστα ε, ελάχιστη πυγμή. Οι αποφάσει τη δεν είναι αποτελεσματικέ. Πώληση όπλων και ε, αρπαγή των πόρων άλλων λαών. Αυτό κάνει η Ευρώπη. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα γενεσιουργά αίτια και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχει γαλάζια κάρτα του κύριο Βάγγελ. Θέλετε να απαντήσετε. Κύριε Βάγκελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφε. Υπάρχουν συνάδελφοι από την ομάδα σας ε, που ε, προσπαθούν ε, να αξιολογήσουν την κατάσταση. Εγώ θα ακούσω τις τελευταίες σας φράσεις. Συζητάμε σήμερα για την συμφωνία με την Τουρκία και συζητάμε πάρα πολλά θέματα. Ε, καθώς και το κατά πόσο μπορεί να ελέξει μια πολιτική εν της ένταξης μιας χώρας, καθώς και άλλα θέματα. Με βάση τη συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα, ε, νομίζετε ότι ε, δεν θα πρέπει να μιλήσουμε για τα γενεσιουργά αίτια αυτής της κρίσης. Εμείς δεν είμαστε ανθρωπιστική οργάνωση, είμαστε πολιτικοί και θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ουσία και τις αιτίες της καταστροφής στη Μέση Ανατολή. Είμαστε πολιτικοί άντρε και γυναίκε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσει από τη σκοπιά τη πολιτική και τη νομοθεσία. Δεν είμαστε καμία φιλανθρωπική οργάνωση, ούτε ένωση εθελοντών. Πρέπει όμω να δούμε τι λύσει υποβάλλουμε επιτάπητο. Αυτέ που προτείνουμε θα πρέπει να είναι χειροπιαστέ και νομοθετικέ. Όχι προτάσει που έρχονται από μη ανθρωπιστικέ οργανώσει. Εγώ σα μίλησα για ανθρωπιστικού διαδρόμου, για εμπάργκο στην πώληση όπλων σε χώρε που βρισκόνται σε πόλεμη κατάσταση. Μίλησα για νόμιμε διώξει και οδούς πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί, δεν βλέπετε ότι είναι προτάσεις χειροπιαστές που θέλουν να χτυπήσουν ε, τα, τη ρίζα του κακού, τα αίτια των μεταναστευτικών ροών. Γιατί αυτές οι μεταναστευτικέ ροέ, ε, αυτές κατε αυτές, υπήρχαν ανέκαθεν. Ένα πράγμα είναι ο θέλει μετακίνηση των ανθρώπων και άλλο είναι η δίωξη και ο πόλεμος που εξαναγκάζουν τους ανθρώπους να αρχίσουν να διαφεύγουν. Μην γίνουμε συνένοχοι. Ευχαριστούμε ο κύριο Μπέι. Στις 18 του Μαρτίου η καγκελάριο Μέρκελ και άλλοι λεγόμενοι διαπραγματευτές αυτής της συμφωνίας με την Τουρκία υποχώρησαν σε όλες τις απαιτήσεις του Σουλτάνου Ερντοάν. Αιώνια κορόιδα στη νέο, νέο Οθωμανική φάρσα, οι ηγέτες που ε, είναι επικεφαλής των ε, τυχών της ε, Υπήρου μας υπέγραψαν νέα λευκή συμφωνία στον πυρομανή πυροσβέστη Ερντογάν. Του διπλασιάσαμε το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι μα. Παρά τι σκοτεινέ σχέσει των Τούρκων με του βάρβαρου του Ισλαμικού κράτου και ενώ η Τουρκία αφήνει να θησαυρίζουν οι μαφίε των διακινητών, αποφασίσαμε να δώσουμε στα 80 εκατομμύρια των πολιτών τη Τουρκία πρόσβαση χωρί περιορισμού στο, ε, στο χώρο Σέγγεν. Γι' αυτό ο Επίτροπο Αβραμόπουλο μου είπε χθε και μα είπε χθε και παραθέτω ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα εποχή Ανθρώπινη κινητικότητα. Τον επόμενο Ιούλιο, την 1η Ιουλίου, η Σλοβακία θα αρχίσει να προεδρεύει στην Ένωση. Ο Πρωθυπουργό τη Σλοβακία, ο Ρόμπερτ Φίκο, καταγγέλει αυτό που αποκαλεί τελετουργική αυτοκτονία της Ευρώπης. Όπως και οι Ούγγροι, Πολωνοί και τέχοι συνάδελφοί του βλέπει ότι η πολυπολιτιστική ουτοπία σας είναι αποτυχία. Ο κύριος Επιτίδιος. Παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε η συμφωνία της ευρωπαϊκής ενώσεως με την τουρκία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος αυτή είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. καταρχάς η τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λαθρέας διακινήσεως ατόμων από το έδαφος της προς την ελλάδα. τα πλοιάρια τα οποία μεταφέρουν τους παράνομους μετανάστες από την τουρκία στην ελλάδα ξεκινούν πολύ νωρίς το πρωί. η τουρκική ακτοφυλακή αρχίζει τις περιπολίες στι 11 το πρωί. το ίδιο κάνουν και τα πλοία του νατο πώς είναι δυνατόν να εντοπιστούν τα πλοιάρια των παρανόμων ε, διακινητών. επιπλέον η τουρκία έχει χορηγήσει μεγάλο αριθμό εκατοντάδων χιλιάδων πλαστών συριακών διαβατηρίων σε αφγανούς και Πακιστανού. αυτοί όταν επαναπροωθηθούν στην τουρκία οι τουρκικές αρχές εύκολα θα διαπιστώσουν ότι τα διαβατήρια είναι πλαστά αφού αυτοί τους τα έχουν χορηγήσει και θα τους επαναπροωθήσουν στην ελλάδα. άρα λοιπόν αυτοί θα μείνουν εκεί και θα υπάρχει πρόβλημα. Τέλο, υπάρχει πληροφορία αλλά και η βεβαιότητα ότι οι παράνομοι μετανάστες θα αρνηθούν ότι η τουρκία είναι χώρα ε, ασφαλής και δεν θα θελήσουν να πάνε εκεί όπου θα μείνουν στην ελλάδα. ας αφήσετε λοιπόν τις υποκρισίες και ας πιέσετε την τουρκία να εφαρμόσει τη συμφωνία. διαφορετικά ο εξαθλιωμένος από τα μνημόνια ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει στην κυβέρνησή του να εγκρίνει τη χρηματοδότηση με τρία δισεκατομμύρια ευρώ της τουρκίας. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου, η συζήτηση αυτή δημιουργεί μεγάλη συγκίνηση. Γιατί γνωρίζουμε και τα προηγούμενα πριν από την Σύνοδο του Μαρτίου. Ξέρουμε γιατί χρειαζόμαστε τη συμφωνία αυτή. Διότι διακινδυνεύουμε να χάσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων. διατρέχαμε τον κίνδυνο επανεισαγωγή εσωτερικών ελέγχων, ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Όλοι ξέρουμε ότι η συμφωνία με την Τουρκία είναι αποτέλεσμα λεπτών συμβιβασμών και γνωρίζουμε ποια είναι τα νομικά προβλήματα και οι προκλήσεις. Παρ' όλα αυτά η συμφωνία αυτή αποτελεί πραγματική βοήθεια προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία οι παρούσες συνθήκες ε, δεν έχουν προηγούμενο και γι' αυτό και τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να είναι μέτρα που δεν έχουν ληφθεί στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να λησμονήσει τις ε, κοινέ της αξίες. Μετά τη διάσκεψη κορυφής στη Μάλτα στις 11 Νοεμβρίου και μετά τη συμφωνία με την Τουρκία, ε, βλέπω ότι σιγά σιγά υπάρχει συμφωνία και με άλλες χώρες διότι η διεθνής προσέγγιση είναι η μόνη λύση. Χαιρετίζω τα μέτρα για τη χαλιβουργία γιατί πρόκειται για 300.000 θέσεις εργασίας, ε, καθώς και πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας έμεσα και είναι κάτι το οποίο αφορά την ε, χώρα μου, την Πολωνία ενώ παράλληλα έχουμε και μια δύσκολη κατάσταση στην αγορά της γεωργίας και ιδιαίτερα στο γαλακτοκομικό τομέα. Ο ενεργειακός εφοδιασμός ε, με αέριο και οι διεθνείς συμφωνίες για την ενέργεια και η διαφάνεια είναι σημαντικό θέμα. Ο κύριος, Ο κύριος Αγαπητοί συνάδελφοι, μα συμφωνούμε. Η συμφωνία με την Τουρκία είναι μόνο τμήμα της λύσης. Η Τουρκία για θέματα μετανάστευσης και προσφύγων είναι σημαντικός εταίρος μας. Αλλά η βασική ευθύνη είναι δική μας, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες, με ευρία πλειοψηφία, εγκρίναμε μια έκθεση πρωτοβουλία που καθιστά σαφές τι επιδιώκουμε. Θέλουμε περισσότερη ενδοευρωπαϊκή αλληλεγγύη, θέλουμε περισσότερες νόμιμες δυνατότητες μετανάστευσης, θέλουμε η διαδικασία του Δουβλίνου να επανεξεταστεί, θέλουμε να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του Σέγγεν. Και θεωρώ ότι αυτά είναι οι προτεραιότητές μας, όπως και πριν. Η συμφωνία για την Τουρκία μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο αν υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Άρα είναι και θέμα διαχείρισης. Πρέπει λοιπόν να λειτουργήσουμε πολύ συγκεκριμένα, να υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες. Αν δεν μπορώ να υποβάλω αίτηση ασύλου, δεν μπορώ να επιστραφώ. Άρα το θέμα είναι πώς θα στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές. Και με λυπεί αγαπητέ Γκραφ Λάνσδορφ το ότι πάντα διαμαρτυρόμεθα για τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Ε, απευθύνομαι στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δεν μπορεί από τις 30.000 υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθήσει και αυτός με κάποιους Να το βοηθήσω και εγώ ίδιο άμα χρειαστεί. Και τελευταίο. Χρειαζόμαστε ρεαλιστικές λύσεις. Οι εικόνες που βλέπουμε στην ειδομένη είναι απαράδεκτες. Πρέπει να δράσουμε λοιπόν. Και μετά να δει για τις επιπτώσεις του δικαίου. Πρόεδρος, πρέπει να είμαι λίγο πιο αυστηρή με το χρόνο ομιλίας. Υπάρχει μπλε κάρτα από τον κύριο Ρόπε. Τη δέχεστε? Από τον κύριο Ρούπε. Τη δέχεστε, ωραία. 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Θέλω να θέσω ένα θέμα για τις δικαιολογίες των κρατών μελών. Οι επάλληλοι μας ε, επισκέφθηκαν ε, τους ε, καταβλημούς και ρώτησαν και κανένας πρόσφυγος δεν θέλει να έρθει στις βαλτικές χώρες. Θεωρείτε ότι πρέπει να τους υποχρεώσουμε να έρθουν στις βαλτικές χώρες. Ο κύριος Φλέκενστάιν. Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσουν αυτά που λέτε για καταναγκασμό. Δεν είναι θέμα να καταναγκάσουμε πρόσφυγες. Έχουμε 28 κράτη-μέλη. Αυτό είναι το θέμα. Και συμφωνήσαμε να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το θέμα δεν είναι να υποφελούμεθα μόνο από τα θετικά και να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες και για τη Γερμανία. Και εμείς δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά Αλλά αυτό καλεί πάντα να γίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλληλεγγύη είναι διπλή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ, συνεχίζει η Πρόεδρο. Ένα λεπτό η κυρία Τρεμπέσιου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στη διάσκεψη κορυφή το Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν πίεση τη Γερμανία έκανε αυτή τη συμφωνία με την ε, Τουρκία ε, ε, ελπίζει η κυρία Μέρκελ ότι τώρα η Τουρκία θα εμποδίσει τη ροή των ε, προσφύγων. Έκτοτε η Γερμανία στα μέσα ενημέρωσης ζει μια νέα εποχή με τον πρόεδρο Ερντογάν και φαίνεται ότι η καριέρα της κυρίας Μέρκελ αυτή τη στιγμή εξαρτάται από τον κύριο Ερντογάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την προστασία των εξωτερικών της συνόρων μόνη της και θα πρέπει να δώσουμε το σήμα ότι η Ευρώπη μπορεί να δράσει με τη δική της δύναμη. Αυτό θα πρέπει να τονίσουμε και δεν θα πρέπει να υποκύπτουμε σε ε, ε, συμβιβασμούς. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να φροντίσουμε τις περιφέρειές μας καλύτερα. Θα πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι από την Τουρκία και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και με την Ιορδανία και το Λίβανο. Ευχαριστούμε κυρία Ίντεφελ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βεβαίως και πρέπει να διαπραγματευόμαστε ε, με τις ε, γειτονικές μας χώρες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αναθέτουμε τις ευθύνες για τα δικά μας προβλήματα. Θέλουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο ισότιμων εταίρων. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδύναμη αφού δεν επιλύουμε τα δικά μας προβλήματα και οι Τούρκοι το συνειδητοποιούν αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε μάθει από τις προηγούμενες εμπειρίες μας όπως το 2010 όταν διαπραγματευτήκαμε συμφωνία με τον κύριο Καντάφη για να κρατάει τους πρόσφυγες εκεί. Και τότε θυμόμαστε τι επιτυχίες είχαμε άκουσα ομιλητέ εδώ να λένε νωρίτερα ότι κύριε Τούσκ, recht ε, in ordnung είναι το σωστό αυτό που συνέβη. Αλλά δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι εγώ. Ακούμε ιστορίε ανθρώπων που ξαναστένονται στη Συρία με ε, μηδέν απάντηση από το Συμβούλιο και τα κάτι μέλη για αυτέ τι περιπτώσει. Αυτό το βρίσκω όνειδος. Η Ήπειρος αυτή, η πλουσιότερη, η πλέον ευημερούσα και οι ελευθερότεροι στον κόσμο τα ανέχεται αυτά. Και δεν μπορούμε να δώσουμε καμία απόκριση στην κατάσταση αυτή. Και εν τέλει, αυτέ τι μέρε τα λέμε και ξανά και ξανά για τι αξίε μα, τι δικέ μα τι αξίε, πώ οι πρόσφυγε πρέπει να τι ενστερνιστούν. Ε, α τι κρατήσουμε επιτέλου ψηλά αυτέ τι αξίε και α φροντίσουμε να έχουν κάτι να σεβαστούν και να ακολουθήσουν αυτοί οι πρόσφυγε. Ε, με συγχωρείτε, πρέπει να σα διακόψω, γιατί θέλω να με όλου ε, για το χρόνο του. Ο κ. Παπαδημούλη. Βέμπερ, σταματήστε αφήστε επιτέλους να αδικείτε και να προσβάλλετε και την ελλάδα αλλά και την αλήθεια. ο κύριος ερντογάν φυλακίζει δημοσιογράφους κλείνει εφημερίδες δεν εφαρμόζει καν τη συμφωνία αλλά εσείς τον χαϊδεύετε και κατηγορείτε τον τσίπρα. ο κύριος όρμπαν ο ακροδεξιός δεν δέχεται ούτε έναν πρόσφυγα στην ουγγαρία αλλά εσείς τον χαϊδεύετε γιατί είναι στην ομάδα σας και φυσικά πάλι καταγγέλλετε τον Τσίπρα. Ίσως να τον βλέπετε και στον ύπνο σας. Ο ελληνικός λαός είναι υπερήφανος με μεγάλη ιστορία και προσφορά και δεν ανέχεται αυτές τις προσβολές του κάθε κύριου Βέμπερ. Κύριε Τούσκ και κύριε Γιούνκερ, ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι φορτώσατε την αποτυχία τη δική σας να εφαρμόσετε τις αποφάσεις του σεπτεμβρίου για αναλογική μετεγκατάσταση στους ώμους ενός κράτους μέλους της ελλάδας εξοραίζοντας παράλληλα την τουρκία. η χώρα μου η ελλάδα σηκώνει ένα τεράστιο βάρος εξαιτίας του πολέμου της γεωγραφίας αλλά και της ευρωπαϊκής αποτυχίας και ο ελληνικός λαός χρειάζεται περισσότερη βοήθεια και αλληλεγγύη όχι να χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος τράγος ή ως σάκος του μπόξ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν αρχίζουμε να ε, κλείνουμε τους ανθρώπους σε περιορισμένους χώρους, θα πρέπει κάτι να σκεφτούμε να κάνουμε και για να τους βρούμε φαγητό, να τους βοηθήσουμε, να τους προσθέσουμε τα παιδιά τους. 28 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Τι έκαναν, κατέληξαν σε μια συμφωνία με την Τουρκία και δεν τα έλαβαν αυτά υπόψη τους. Δεν φαίνεται να έχουν προβλέψει τι θα γίνει. Ε, δεν φαίνεται να σκέφτηκαν τι θα γίνει με τη διατροφή των ανθρώπων αυτών, με τα παιδιά τους, με την προστασία τους. Δεν φαίνεται να υπάρχουν δικηγόροι. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα κάνουν κάποιο βήμα για να υλοποιήσουν άραγε αυτή τη συμφωνία. Και θα πρέπει ενδεχομένως να στραφούμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Μόνοι μας δεν γίνεται νέα κορίτσια 14 ετών να είναι κλειδωμένα μαζί με άνδρες ενήλικους σε ένα κέντρο κράτησης. Με συγχωρείτε, αλλά θέλουμε, αν μπορείτε να δεχτείτε γαλάζια κάρτα την κυρία Γιάτεν Μάκη. Τη δέχεστε? Ακούστε, ε, πολλοί είναι αυτοί που εδώ έχουν ε, επικρίνει τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Δεν είναι τέλεια, αλλά έχουμε καμία εναλλακτική. Τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώστε μου εσείς μία άλλη εναλλακτική λύση. Τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κάτι μέλη της. Η κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για κοιτάξτε, έχω ένα ε, σχέδιο όλη την ε, επαναγκατάσταση από τις τρίτες χώρες με νόμιμη ε, πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους. Δεν είναι το θέμα τι κάνει Ερντογάν και Τουρκία. Δεν μίλησα γι' αυτό. Είπα τι δεν κάνουμε εμείς. Εμείς τι παραλείπουμε. Και εμείς δεν φροντίζουμε καν αυτούς που έχουμε κλεισμένους σε κέντρα κράτησης. Αυτό λέω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάξας, 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει περάσει ένας μήνας από την συνάντηση κορυφής. Μικρό χρονικό διάστημα, αλλά επαρκές για να δούμε τις τάσεις που διαγράφονται. Με βάση αυτή τη συμφωνία, κάποιες εκατοντάδες παράνομων μεταναστών ε, επεστράφησαν. και κάποιοι πρόσφυγες ε, έγιναν δεκτοί στην Ευρώπη. Η τσεχική δημοκρατία είναι κατά των ποσοστώσεων κατανομής. Άρα συνολικά οι εξελίξεις δεν είναι θετικές. Κάπως ε, δημιουργήσαμε ένα μηχανισμό ελέγχου, αλλά δεν έχουμε λύσει καθόλου το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε θαραλέες αποφάσεις. Τα εξωτερικά μας σύνορα πρέπει να προστατευτούν. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε καθόλου παράτυπη μετανάστευση. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να δεχθούν τέτοια πράγματα. Πρέπει να μην εφαρμοστούν οι ποσοστώσεις κατανομής. Το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευση μπορεί να δημιουργήσει και οικονομικά προβλήματα. Το πρόγραμμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εφαρμοστεί τάχιστα με συγκεκριμένα μέτρα ούτω ώστε να γίνει πραγματικότητα το πρόγραμμα αυτό για να επιληθούν τα οικονομικά προβλήματα που συσσωρεύονται και δεν αντιμετωπίζονται. Τα κράτη-μέλη πρέπει να δείξουν περισσότερη να αποκτήσουν καλύτερα περισσότερη ευελιξία για, την, για τον καθορισμό των συντελεστών του ΦΠΑ. Και έτσι μόνο θα βοηθήσουμε την κατανάλωση γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαλβίνη, ευχαριστώ πρόεδρε. Πολλαπλή συζήτηση, πολλαπλή απόδειξη ότι η Ευρώπη δεν υπάρχει. Η Ευρώπη επικοδομήθηκε σε ένα λανθασμένο νόμισμα και τώρα πεθαίνει λόγω της μετανάστευσης. Κάποιος ε, αποφάσισε να φέρει μερικά εκατομμύρια σκλάβους και εδώ σε αυτό το μέγαρο μιλάμε για μεταναστεύσεις και ε, τη συμφωνία με την Τουρκία με τόσα δις ε, ευρώ. Την Τουρκία που αρνείται τη γενοκτονία των, του 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων ε, που κατέχει στρατιωτικά το έδαφος ενός κυρίαρχου κράτους μέλους που συμμετέχει σε αυτόν τον οίκο που θέλει να μπει στην Ευρώπη και με ε, με, παρα, παραχαράσοντας την ευρωπαϊκή ιστορία και την εμπειρία μας και την πορεία μας. Εδώ μιλάμε για τρέλες και ανοησίες, ενώ ε, αποβιβάζονται 3.000 λαθρομετανάστες από τις αρχές του χρόνου στην Ιταλία και στις ακτές της, το διπλό από πέρσι, και 5% είναι το σύνολο. Λοιπόν, τι είναι αυτή η Ευρώπη. Ευχαρίστω να φύγουμε από αυτήν, αν θέλετε, νομίζω, αν θέλετε να μα πείσετε εμένα και του 20 εκατομμυρίου ανέργου με του οποίου κανεί δεν ασχολείται, ότι αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Ευχαριστούμε ο κ. Παπαδάκη για 1,5 λεπτό. Βρίσκεται στην αίθουσα. Ναι, ευχαριστώ. Η απόφαση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία ρίχνει νέο λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων με ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην επέμβαση στη Συρία η απόφαση να ανοίξει ακόμα ένα κεφάλαιο για την ένταξη της τουρκίας στην ευρωπαϊκή ένωση επιβραβεύει και νομιμοποιεί την αυξανόμενη επιθετικότητα της αστικής τάξης της τουρκίας σε συρία αιγαίο και κύπρο. για ποια αλληλεγγύη μιλάτε στους πρόσφυγες με φράχτες φυλακίσεις απελάσεις και απαράδεκτο πινκ πονγκ προσφύγων; όλα επιβεβαιώνουν ότι επιχειρείτε να αντικαταστήσετε τη συνθήκη της γενέβης ό,τι δηλαδή έχει μείνει όρθιο από την προστασία των προσφύγων με απάνθρωπους ευρωνοσιακού μηχανισμούς. κύριε βέμπερ γιατί σκόπιμα μπερδεύετε τις πολιτικές ταυτότητες και μιλάτε δήθεν για κομμουνιστές του σύριζα αναζητώντας κιάχτρο. ο σύριζα είναι η νέα σοσιαλδημοκρατία στην ελλάδα στηρίζει το μεγάλο κεφάλαιο προωθεί βάρβαρα δεργατικά μέτρα και μνημόνια όπως και άλλωστε και τα σοσιαλδημοκρατικά και φιλελεύθερα κόμματα κάνει εκκλήσεις για να υλοποιηθούν οι απαράδεκτες αποφάσεις της ευρωπαϊκής ένωσης και το προσφυγικό αλλά και λέει για την αποτελεσματική δράση του νατο και άγχεται για την αποτελεσματική δράση του νατο στο αιγαίο. το κομμουνιστικό κόμμα της ελλάδας καλεί το λαό αποφασιστικά να οργανώσει την πάλη του με 48 ώρια απεργία μπροστά στα νέα βάρβαρα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση σύριζα ανέλ που πλήττουν συνολικά και τον ελληνικό λαό και τους πρόσφυγες. Και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα τέλη του 2015 θυμάμαι ο πρόεδρος Γιούγκερ μας είχε πει ότι ήταν επίγον να βρεθεί μια λύση πριν από την Άνοιξη και πριν αρχίσουν να αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές η συμφωνία με την Τουρκία τουλάχιστον υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε, διότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι το ορίζει η Τουρκία και χρησιμοποιεί την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να βρεθεί κανείς σε επιτόπου για να δει πόσο δεν λειτουργούν τα πράγματα και πόσες ελλείψεις υπάρχουν στη διαδικασία ασύλου στην Αθήνα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια έκρηξη των αιτήσεων ασύλου με 500.000 μετανάστες και υπάρχει ε, έλλειψη προσωπικού επιτόπου και από τα κράτη-μέλη η βοήθεια που ε, έχει υποσχεθεί δεν φτάνει. Δεν πρέπει να είμαστε ε, αφελείς. Ο πρόεδρος Ερδογάν υπενθυμίζει με χαρά ότι η Τουρκία δεν θα τηρήσει το δικό της μέρος της συμφωνίας αν δεν τηρήσει τις υποσχέσεις της η Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια αναφέρεται στις θεωρήσεις διαβατηρίου που βιαστήκαμε να υποσχεθούμε στους Τούρκους. Πολλοί Ευρωπαίοι ε, αποφεύγουν να αναλάβουν τις ευθύνες της και η Γαλλία ε, δεν αναλαμβάνει να κινητοποιηθεί και άφησε την κυρία Μέρκελ να διαπραγματευτεί μόνη της με την Τουρκία. Δεν θα πρέπει μέσα σε όλα αυτά να ξεχνάμε και μια άλλη κατεπίγουσα ανάγκη, το να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και να προωθήσουμε την απασχόληση. Και εδώ θέλω να μιλήσω για την χαλιβουργία. Δεν θέλουμε να προστατεύσουμε μια βιομηχανία που παραπέει, αλλά να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε τη βιομηχανία του να αντιμετωπίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό, να αντιμετωπίσει ε, το dumping και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα σύντομα. Ευχαριστώ. Κύριε Ροντρίγκε, ένα μισή λεπτό. We Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η συμφωνία με την Τουρκία είναι μια προσωρινή και αντιφατική λύση. Αυτό που χρειαζόμαστε στην πράξη είναι ευρωπαϊκά ε, μέσα τα οποία θα μας βοηθήσουν να ανακτήσουμε έλεγχο της κατάστασης ε, με τα σωστά πρότυπα. Ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να θέσουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες ε, ε, οι πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής ε, προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες ασύλου θα τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεύτερον, θα πρέπει να μην δημιουργηθούν γκέτο μέσα στις πόλεις μας για λόγους κοινωνικής συνοχής και για λόγους ασφαλείας, για να αποφύγουμε κινδύνους για την ασφάλεια. Τέλος, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό σύστημα συνόρων για την Ευρώπη, όχι η Χθε και όχι τύχη, αλλά ένα δίκτυο ε, συνόρων που θα βοηθήσει, θα βοηθήσει τους ε, ε, πληθυσμούς της Ευρώπης σύμφωνα με τα όσα έχουν αποφασίσει οι ευρωπαϊκές αρχές. Η ευρωπαϊκή κυριαρχία είναι αυτό το οποίο διατρέχει κίνδυνο αυτή τη στιγμή, γιατί η ευρωπαϊκή κυριαρχία είναι μια ισχυρή έννοια και οι πολίτες κατανοούν ότι πρέπει να περάσουμε σε μια νέα φάση όπου θα δημιουργήσουμε ε, τις βάσεις για να έχουμε την κυριαρχία ε, επί των πόρων μας, επί των συνόρων μας και επί των προτύπων ε, που έχουμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι λοιπόν το μέλλον για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χαλαγό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, λέγεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και παραθέτω ότι πολλά στοιχεία τη κοινή ευρωπαϊκή απόκριση στην κρίση των μεταναστών ήδη έχουν ε, λειτουργήσει σήμερα και δίνουν αποτελέσματα. Τέλο παραθέματο. Πολύ αισιόδοξη δήλωση. Τα κοινά μα μέτρα, όπω το σύστημα επαναγκατάσταση, δεν έχουν λειτουργήσει καθόλου τώρα και μάλλον οι μονομερείς αποφάσεις που λαμβάνουν τα επιμέρους κρατημέλη έχουν μειώσει τη ροή μεταναστών ή κάπως την έχουν κατευθύνει αλλού. Αναφέρομαι όλος ιδιαίτερος στην ε, επαναφορά των συνοριακών ελέγχων και της ε, λήψης μονομερών αποφάσεων για κλείσιμο των συνόρων σε επίπεδο κρατών μελών. Εδώ αυτό είναι απαράδεκτο ε, ως προς την εξέταση των ε, τήσεων άνθρωπων που έρχονται από την Τουρκία. Και ήδη διαρωτώ με τι γίνεται εντός των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό κύριο Στελίτσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Τούσκ, πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι τα σχόλιά σα για τη συμφωνία με την Τουρκία, ιδίω τι επεκτητικές σα παρατηρήσει, αλλά θα είχα και μια ερώτηση. Πώ παρακολουθούμε και ελέγχουμε την υλοποίηση της τουρκικής πλευράς, Τη συμφωνίας από την τουρκική πλευρά. Πώς αποτιμούμε την συμφωνία και σε τι πορίσματα μπορούμε να καταλήξουμε. Κύριε Γιούνκερ, δύο παρατηρήσεις. Για το θέμα της μετανάστευσης. Ζητήσατε καθοδήγηση από τις πολιτικές ομάδες. Δικαίως. Θα έλεγα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμπεριέχει χρήσιμα και αποτελεσματικά στοιχεία κάμποσα τέτοια. Θα βασιζόμουν σε αυτά. Σε αυτά που θα μπορούσαμε αμελητή και ε, αποτελεσματικά να εφαρμόσουμε και γύρω από τα οποία μπορεί να ε, συνασπιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια παρατηρήση για την Κίνα. Δίκαιο εμπόριο, δίκαιο ανταγωνισμό, αλλά δεν είναι αυτό η Κίνα. Ούτε η χαλιβουργία, ούτε η συσκευασία τη, ούτε σε άλλε ε, σε άλλες εταιρείε και επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Α δράσουμε λίγο πιο γρήγορα και με περισσότερη πυγμή. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό, κύριο Σκουντή. Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης και ε, τουρκίας αποτελεί μαύρη σελίδα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ένωσης και είναι ντροπή σε όσους την έχουν συνυπογράψει. η ευρωπαϊκή ένωση προκειμένου να ξεφορτωθεί από τις πλάτες της ένα πρόβλημα για το οποίο είναι συνυπεύθυνη βάφτισε την τουρκία ασφαλή χώρα αγνοώντας προκλητικά ότι καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. η συνθήκη της γενέβης πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Χιλιάδε πρόσφυγε έχουν εγκλωβιστεί στην ελλάδα χωρί να του δίδεται ουσιαστικά το δικαίωμα ασύλου στη χώρα που επιθυμούν. η αστυνομία τη φύρομ ε, καταπατά τα δικαιώματα των προσφύγων και χρησιμοποιεί ομή βία. η συμφωνία άνοιξε κεφάλαια για την ένταξη τη Τουρκία στην ευρώπη ενώ την ίδια ώρα αμφισβητούνται εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα τη Ελλάδα, καθημερινά παραβιάζεται ο ελληνικό εναέριο χώρο και δημιουργούνται ή επιχειρείται να δημιουργηθούν τετελεσμένα και γκρίζε ζώνε στο αιγαίο με τον νατο παρόν. κύριε σας ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε είναι μετέτρεψε την ηγεσία της ευρωπαϊκής ένωσης σε κομπάρσο σε ένα θεατρικό έργο για την προσφυγική κρίση με πρωταγωνιστή τον κύριο ερντογάν. σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, Πρόεδρε της Επιτροπής, αυτή η συμφωνία με την Τουρκία δεν αποτελεί λύση. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι επιστρέφουμε πρόσφυγες στην Τουρκία και η Τουρκία τους ξαναστέλνει στη Συρία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό που κάνουμε είναι ότι αποποιούμεθα τις ευθύνες μας και αυτό δεν συνάδει με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το οποίο λέει και η Διεθνής Αμνηστία και θα πρέπει να οργανώσουμε αποστολή εκπροσώπων ε, πολιτικής και της κοινωνία των πολιτών για να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει στην πράξη, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Χρειαζόμαστε μια νόμιμη διαδικασία για την επανεγκατάσταση και θα πρέπει ε, όλοι και λέω όλοι και τα κράτη-μέλη που λένε ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην επανεγκατάσταση όλοι θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και όλοι θα πρέπει να δεχθούμε και να υποδεχθούμε ε, πρόσφυγες ε, δεν θέλω να μιλήσω ε, για τα όσα έχουν γίνει στην Αυστρία τις τελευταίες μέρες, αλλά το κλείσιμο του περάσματος του, του Μπρένερ ε, είναι κάτι το, το οποίο είναι αδιανόητο. Θα πρέπει και σε σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνει ανοιχτό και αυτό το σύνορο και όλα τα σύνορα. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λούντγκεν για ένα λεπτό, θα, δεν θα μπορούμε να δεχθούμε άλλε γαλάζιε κάρτε γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Ελπίζω να δείξετε κατανόηση, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε εγκαίρω αυτή τη συνεδρίαση. Ο κύριο Λούντγκεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει με όλες μας τις πολιτικές να προστατεύουμε και τα εθνικά συμφέροντα και γι' αυτό θα μιλήσω εδώ όχι μόνο Ευρωπαίος αλλά κυρίως Σουηδός. Ε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν δέχομαι να προσπαθούμε να επιβάλλουμε το οτιδήποτε στη Σουηδία σαν να ήμασταν υποτελεί σε κάποια υπερδύναμη. με τόσε πιέσει. Η Τουρκία είναι μια χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δεν σέβεται την ε, ελευθερία τη έκφραση. Και παρόλα αυτά παίρνει ένα σωρό χρήματα από του φορολογουμένου του δικού μα. Δεν είναι καν ευρωπαϊκή χώρα η Τουρκία. Ασιατική είναι. Ε, κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να επιβληθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μια πολιτική που οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό ο κύριος Ντεγκράφ. Sorry, could you please put on your Με συγχωρείτε, μπορείτε να ανοίξετε το μικροφωνό σας. Πρόεδρε, η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων ε, για την Τουρκία η επιστροφή των προσφύγων από την Τουρκία στη Συρία, αυτή είναι η συμφωνία που πετύχαμε. Και τι κάνει η Τουρκία, ε, δεν αφήνει σε ησυχία τους Κούρδους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους πολίτες της. Δεν γίνονται σεβαστά τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά γίνονται αποδεκτά μόνο και μόνο για μια συμφωνία αυτού του είδους. Υπάρχει πρόβλημα ηθικής από την πλευρά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά μπουχτίσαμε. Φτάνει. Δεν μπορούμε να αντιδράμε έτσι, να κλείνουμε απλώ τα σύνορα και να στέλνουμε πίσω του μετανάστε κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ για 1,5 λεπτό ο κ. Γκοτσάλε Πόν. Είναι πολύ εύκολο να είναι κανεί υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν τα προβλήματα είναι στην άλλη άκρη τη Μεσογείου. Είναι πολύ πιο δύσκολο όταν είναι μπροστά μα. Είναι σαφέ ότι οι πρόσφυγοι πρέπει, οι πρόσφυγες, συγγνώμη, πρέπει να ε, υφίστανται σωστές διαδικασίες αλλά μοιάζει να μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι διαδικασίες παρά τα άτομα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα η Γερμανία και η Ελλάδα πρέπει να τα κάνουν όλα οι εχθροί της Ευρώπης δεν είναι αυτοί που διασχίζουν ε, τις ε, θάλασσές μας με αυτά τα φουσκωτά ούτε αυτοί που πνίγονται οι εχθροί είναι αυτοί που σπρώχνουν τους πρόσφυγες προς τα σύνορά μας και αυτοί που χαμογελούν όταν οι Ευρωπαίοι παραβιάζουν τις αρχές τους. Οι εχθροί της Ευρώπης είναι αυτοί που προκαλούν την τρομοκρατία, όχι αυτοί που διαφεύγουν, προσπαθούν να αποφύγουν την τρομοκρατία. Η Τουρκία βεβαίω είναι μέρο τη λύση, αλλά η Τουρκία δεν είναι η λύση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μια υπηρεσία που μπορούμε να την αγοράσουμε με ευρώ ή τα πιστεύουν και τα εφαρμόζουν ή όχι. Και δεν θα σταματήσει η κρίση αν κλείσουμε την πόρτα στου ε, φτωχού Σύρου και την ανοίξουμε για τους πλούσιους Τούρκους ούτε αν δώσουμε ως υπεργολαβία σε κάποιους την διαχείριση της κρίσης συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Έχει μία τιμή λοιπόν η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν έρθει η ώρα πρέπει να είναι κανείς υπέρ της Ευρώπης και πρέπει να αποδείξει την αλληλεγγύη του και για να δίνει κανείς μαθήματα πρέπει στην πράξη να τηρεί αυτά τα οποία διακηρύσει. Και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν μπορεί να δώσει μαθήματα ούτε για την προστασία των ε, φτωχών και διοκομένων. Πρέπει πολλά να μάθουμε ε, και πρέπει να ξεκινήσουμε την εργασία της Κομισιόν. Ευχαριστώ όλοι, Πρόεδρος. Ενάμιση λεπτό. Η κυρία Γκυγιώμα. Ευχαριστώ. Η συμφωνία με την Τουρκία είναι ικανοποιητική. Η απάντηση είναι όχι. Ε, και προσπάθησε να το τυλίξουν σε ένα ωραίο πακέτο όλο αυτό το πακέτο της συμφωνίας και ίσως ε, ε, να φαίνεται ότι συνάδει προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο αλλά στην πράξη η απάντηση είναι αρνητική. Δεν είμαι η πρώτη που το λέω, είναι πολλοί οι άλλοι συνάδελφοι που το είπαν ότι η επιστροφή των προσφύγων προς την Τουρκία δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με τα δικαιώματα ασύλου και η όλη η συμφωνία δεν είναι ικανοποιητική. Οι δικαστές θα πρέπει να αποφασίζουν ε, για ε, ε, την ορθότητα της συμφωνίας, αλλά προς το παρόν αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η συμφωνία δεν είναι καλή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα πρακτικής ρύθμισης, πρακτικών ρυθμίσεων στην Ελλάδα για να μπορέσει να λειτουργήσει η συμφωνία και η συμφωνία δεν φαίνεται να μπορεί να εφαρμοστεί όπως περιγράφεται στα χαρτιά και αν καταφέρουμε να εμποδίσουμε με οποιοδήποτε τίμημα τους πρόσφυγες να περνάνε στο Αιγαίο, αυτοί θα βρουν άλλες οδούς προς την Ιταλία ή αλλού. Πρόκειται για μια για ε, ένα φρικτό κατασκεύασμα που σιγά σιγά θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα. Ε, τις κριτικές που ακούγονται πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά. Έχω πολλές επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Είναι ε, επικίνδυνη αυτή η συμφωνία. Δεν μπορέσαμε να διαμορφώσουμε μια εναλλακτική πρόταση γιατί δεν υπάρχει αλληλεγγύη εκ μέρους των κρατών μελών. Ένα λεπτό, κύριος Βαντάλεν. Ε, πρόεδρε, η συμφωνία αυτή ε, με την Τουρκία είναι σαν να δούρει ο που έρχεται από την Τουρκία. Το αντικείμενο είναι κάποιες εκατοντάδες πρόσφυγες να γυρίσουν από την ε, Ελλάδα προς την Τουρκία και κάποιοι από την Τουρκία προς άλλες χώρες, ενώ στην Ιταλία έρχονται τώρα χιλιάδες κάθε μέρα. Απελευθερώνουμε τις θεωρήσεις διαβατηρίου για τους Τούρκους που θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με γίνονται προτάσεις και για ένταξη της Τουρκίας και τελικά τι επιτυχάνουμε. Η ομάδα Juncker Timmermans έχει χάσει την εμπιστοσύνη της πέντε μέρες μετά το δημοψήφισμα ε, για την Ουκρανία στην ε, Ολλανδία. Ε, προτείνουμε απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίου. Αυτό πώς μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Πρέπει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, να μας προτείνουν ένα πρόγραμμα με διαδικασίες επιλογής στα λιμάνια για να μπορέσουμε να επιλέγουμε αυτού που είναι πραγματικοί πραγματικά πρόσφυγοι. Κυρία Ντεσάρνες, ένα λεπτό. Βεβαίω πρέπει να υπάρξει διάλογο με την Τουρκία για να σταματήσει τουλάχιστον αυτή η τρομερή δραστηριότητα των εγκληματιών διακινητών. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μα κάνει να αποφύγουμε τι δικέ μα ευθύνε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αναθέσει την άσκηση του δικαιώματο ασύλου στι χώρε που την ε, περιβάλλουν. Πρέπει επιτέλου να αναθεωρηθεί το Δουβλίνο, να αρμονίσουμε τι διατάξει μα και να υπάρξουν ασφαλεί δυνατότητε εισόδου για του Σύρου πρόσφυγε, όπω έκανε για παράδειγμα ο Καναδά. Επιπλέον, η Ευρώπη δεν μπορεί να αναθέσει σε κανέναν τον έλεγχο των συνόρων τη. Πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο σώμα άκτο και σύνοριο φυλάκων και να συντονίσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και για τους πολίτες της. Τέλος, η Ευρώπη δεν μπορεί να αναθέσει τη δυνατότητά της να παίξει όλο στην επίλυση του Συριακού σε κανέναν άλλον. Πρέπει να παίξει πολύ πιο ενεργό ρόλο σε αυτό και να ασκήσει και εδώ πλήρω τι ευθύνε τη, να τι αναλάβει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό η κυρία Μίχελ. Κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. 27 κυβερνήσεις καλούν την Ελλάδα να συμπεριφερθεί σαν να ήταν ασφαλής τρίτη χώρα η Τουρκία οι 27 χώρες και ήταν από την άλλη μεριά όταν διαπιστώνουμε την κατάσταση συνειδωμένη και όταν βλέπουμε από πλευρά της Μακεδονίας να αντιμετωπίζονται με σφαίρες καουτσούκ. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι η συμφωνία που συζητάμε. Παρά το ότι υπάρχει αλληλεγγύη στην Ελλάδα από τους Έλληνες και από ακτιβιστές όλη την Ευρώπη, πρέπει οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να καταδικάσει την αντιμετώπιση των προσφύγων στην Ελλάδα ως παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συμφωνία αυτή έχει δημιουργήσει μια κακή κατάσταση λοιπόν. Μάλλον έχει εδρεώσει την κακή κατάσταση αντί να βελτιώσει την κατάσταση εφαρμόζοντας τη σύμφαση της Γενέβης. Η πολιτική αυτή είναι αποτυχημένη. Άρα πρέπει να αλλάξει. για να μην κλέψουμε από την Ευρώπη ε, το, την ιστορία της και το μέλλον της και την ελπίδα από τους πρόσφυγες. Η Τουρκία δεν είναι μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος. Μέρος του προβλήματος και της Συρίας και των Κούρδων και των προσπαθειών να υπάρξει βιώσιμη λύση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έριξον, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Στη Σουηδία λέμε ότι ε, πάντοτε διατρέχουμε κινδύνους ε, όσα μέτρα προφυλάξεων και αν λάβουμε. Προσπαθούμε να επιλύσουμε την προσφυγική κρίση μέσω μιας συμφωνίας με την Τουρκία. Προσπαθούμε να εμποδίσουμε περαιτέρω ροές τελικά ο οδός των προσφύγων θα αλλάξει και θα περνάει από τη Λιβύη παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με την αιτία των κρίσεων. Γιατί δεν έχουν λειτουργήσει συμφωνίες ούτε και με την Λιβύη. Θα θέλαμε να δούμε τις αιτίες. να γίνει η ίδια η χώρα, να γίνει η Λιβύη μια χώρα που θα λειτουργεί για να μην χρειάζεται να φύγουν οι άνθρωποι το κλείσιμο των συνόρων δεν μπορεί να αποτελέσει ε, λύση. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης από όλους μας. ένα λεπτό. Η Frontex πρέπει να ασχοληθεί με 200.000 μετανάστες που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Πρέπει να, μας, να δούμε κατά πόσον αυτό που λέτε εσείς για συμφωνία με την Τουρκία ως επιτυχία είναι ε, αλήθεια. 300 μετανάστες ε, ε, ήδη στην Ελλάδα αυτές τις μέρες πέρασαν και Υπάρχει ακόμη η λαθρέα διακίνησή τους. Ε, εκατομμύρια πέρσι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα αντιμετωπίσετε το επόμενο τσουνάμι μεταναστών με ελέγχου μόνο στα σύνορα. Είναι ανησυχητικό που η Βρετανική σειροφυλακή αντιδρά τόσο γρήγορα. Ήδη σκάφη περιπολίας, ε, πέντε μόνο από την Βρετανία έχουν σταλεί στην Μεσόγειο. Μια συμβολική χειρονομία που έχει όμως αφήσει ευάλωτα και ανοιχτά τα σύνορα της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα χρήματα των Βρετανών φορολογουμένων τι γίνεται, στέλνονται στην Τουρκία για να πάρουν πίσω τους ε, πρόσφυγες με 18 άτομα που έχουν σταλεί εκεί να εργαστούν για το θέμα αυτό, αφήνοντα τη δική μου χώρα προστάτευτη. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει με όλα αυτά. Μόνο να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε. Ευχαριστούμε για ένα μισή λεπτό, κυρία Καρδίνη. Ευχαριστώ. Επικεντρωνόμαστε στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία. Δικαίω, τι να πω. Αλλά δεν κοιτάζουμε τι θα γίνει με το κλείσιμο τη Ευρώπη που θα έχει σοβαρότερε συνέπειε οι οδοί μετατοπίζονται και εγώ ως Ιταλίδα πρέπει να πω ότι ανησυχώ όλος ιδιαίτερος. Βρισκόμαστε στην εμπροστοφυλακή του προβλήματος αυτού. Υπάρχουν νέες ενδείξεις, νέες οδηγίες δίνονται προς τους μετανάστες και η κατεύθυνση είναι ακριβώς η Ιταλία. Η ιστονομία μας έχει ήδη εντοπίσει πολλές ε, ομάδες που είναι έτοιμες να μετακινηθούν. Έτσι μετατοπίζονται εναλλακτικέ οδές από την Ελλάδα και την Τουρκία προς το νέο μέτωπο, την Μεσόγειο. Και αυτό που μας ενισχύει ακόμη περισσότερο είναι ότι μεταξύ 15 και 19 Μαρτίου 4.000 μετανάστες διαχρονιστήκαν στη Μεσόγειο. Ε, ε, ήδη ε, μας δόθηκαν ενισχύσεις από τις γερμανικές ε, ε μυστικέ υπηρεσίε ότι 18.000 άτομα στι ακτέ τη Λιβύη περιμένουν να περάσουν στην Ιταλία. Όμω, είπατε, εκπρόσωπο μιλά για 450.000 άτομα που είναι έτοιμοι να φύγουν από την Λιβύη προ την Ελλάδα. Μα ανησυχούν πάρα πολύ όλα αυτά. Όπω αυτή η περίοδο αδράνεια που επέτρεψε στα ευρωπαϊκά κράτη να επαναφέρουν του συνοριακού ελέγχου στα σύνορά του. Εάν αυτοί δεν ανακληθούν και αν αυτή η αναστολή του Σέγγεν ε, ή το κλείσιμο των σύνορων διατηρηθεί για ακόμη δύο χρόνια, τι θα γίνει, θα θωρακιστεί προ την Νότια Ευρώπη, η Ευρώπη, η Κεντρική και η Βόρεια. Εδώ λοιπόν απευθύνω έκκληση. Εάν δεν δούμε το μεταναστευτικό συνολικά, η Ευρώπη τελικά αυτή η ίδια θα αναπαγίσει στη Μεσόγειο. Ευχαριστούμε και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Πύρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται η μια την άλλη για να αντιμετωπίσουν τις ανθρωπιστικές υποθέσεις με τρόπο σωστό. Εδώ και χρόνια λέγαμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά όσο Όμω ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας οι εξελίξει. Και δεν φανταζόμαστε ότι τόσοι Σύριοι θα ξεφύγουν προς την ε, ε, ευρωπαϊκή, ε, θα διαφύγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ροή αυτή χιλιάδων ανδρών, γυναικών, παιδιών που δεν μπορούμε να τις συγκρατήσουμε. Δεν έχουμε επιδείξει αρκετή αλληλεγγύη. Συμφωνία με την Τουρκία σίγουρα δεν είναι τέλεια. Σίγουρα δεν δίνει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, όμως είναι τουλάχιστον μια απόπειρα. Είναι μια πρώτη προσπάθεια να εξαλείψουμε αυτά τα χρηματοπλέγματα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποδεχόμαστε αυτό. Πρέπει να προσπιστούμε τις αξίες μας, αλλά πρέπει και με την Τουρκία να μπορούμε να ε, παρακολουθούμε τον σεβασμό των διεθνούς δικαίου από την Τουρκία την ίδια. Ε, δεν πρέπει να στέλνουμε πίσω πρόσφυγες από την Τουρκία στη Συρία, πρέπει να υπάρχουν ε, δυνατότητες ελέγχου και να μην αποστέλλονται πίσω οι Σύριοι στην Συρία από την Τουρκία. Πρέπει οι Ευρωπαίοι φύνοντες να τα δουν όλα αυτά, αποδέχονται μια συμφωνία για την υποδοχή των προσφύγων στην Ελλάδα και για την αποστολή και άλλων προσφύγων προς την Τουρκία χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το τι γίνεται με τους πλέον ευπαθείς πρόσφυγες στο δικό τους έδαφος. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κύριο Σούλικ. Ευχαριστώ πολύ. Οποτεδήποτε έχει επιχειρήσει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινή μας προσέγγιση, η συμφωνία με την Τουρκία, οτιδήποτε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασίζεται πάντα στο ότι οι πρόσφυγες θα διανεμηθούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να αποδεχθεί το γεγονός ότι οι πολίτες πολλών χωρών δεν θέλουν εκατομμύρια μεταναστών στις χώρες τους. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ εκπλήσονται κάθε φορά που οι πολίτες της Ένωσης απορρίπτουν τα μέτρα περαιτέρω ενοποίησης και ψηφίζουν για εξτρεμιστικά κόμματα. Βεβαίω να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, αν τους βοηθήσουμε εκεί που είναι. Δεν θα πρέπει να τους φέρουμε εδώ στις χώρες μας. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Κανείς άλλος δεν θα το κάνει για μας. Σίγουρα όχι η Τουρκία. Αν, αν υπάρχει μια χώρα Σέγγεν που δεν θέλει ή δεν μπορεί να προασπίσει τα σύνορά της θα πρέπει να βγει από το Σέγγεν είτε είναι η Ελλάδα είτε είναι η Ιταλία και θα ε, προστατεύσουμε τα σύνορά μας ε, όπως κάνουμε ήδη στο πέρασμα του Μπρένερ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε η πολιτική μας είναι αυτή η οποία οδηγεί πολλούς να πέσουν τη ζωή τους για να μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο να ζητήσουν άσυλο. θα έπρεπε να είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε πιο ασφαλείς διάβλους για την είσοδο των ε, προσφύγων. Αυτή τη στιγμή θέλει το Συμβούλιο να τιμωρήσει την Ελλάδα επειδή δεν εφαρμόζει σωστά το σύστημα ασύλου αλλά με τρόπο ο οποίος είναι αστυνομικού χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή όμως παραμένει η απόγνωση των ανθρώπων που έχονται στην Ευρώπη φτάνουν στην Ευρώπη πια χωρί καμιά ελπίδα. Αυτοί οι οποίοι θα επιβιώσουν δεν θα ξεχάσουν ποτέ πόσο τους έχουμε κακό μεταχειριστεί. Αυτό σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο κύριε Τούσκ είναι μια ορολογιακή βόμβα για όλου μα. Και δεν θα μειωθεί ο λαϊκισμός αλλά θα αυξηθεί όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Εκ, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια πάρα πολύ λυπηρή και χωρίς ελπίδα εποχή για την Ευρώπη βλέπουμε την αποδόμηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Τουρκία που ουσιαστικά είναι αυτή τη στιγμή αρμόδια για την προστασία της Ευρώπης από τους πρόσφυγες. Η Ευρώπη χάνει την ψυχή της, χάνει την ανθρωπιά της. Πώς μπορούμε εμείς να είμαστε ακόμα υπερήφανοι για την Ευρώπη. Η Τουρκία με τρόπο σαφή έχει παραβιάσει την ε, σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάζει από την άλλη πλευρά. Παρά τις ε, δηλώσεις των οργανώσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ε, θέση των Ηνωμένων Εθνών παραμένει η Ευρώπη σε ένα βρώμικο παζάρι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εξαργυρώνει τη σιωπή της για την πολιτική της Τουρκίας κατά των πολιτών της. Εγώ ως πεπισμένος Ευρωπαίος και ως μέλος αυτού του Κοινοβουλίου πραγματικά νιώθω ντροπή για την αποτυχία μας. Χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική, χρειαζόμαστε μια ανθρώπινη πολιτική, μια πολιτική η οποία δεν θα πρέπει να προδίδει την ευρωπαϊκή ιδέα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριος Μποργέτσιο. Πρόεδρε, η συμφωνία με την Τουρκία έχει πολύ αμφίβολη νομική εγκυρότητα και αυτή η πλειοψηφία που ακούμε να μιλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, που αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει μαζικέ απελάσεις προσφύγων, είναι κάτι που πραγματικά δεν μας αφήνει να είμαστε ήσυχοι. Εδώ ακούσαμε ότι δεν θέλουν να γίνουν κέντρο υποδοχής για τους πρόσφυγες της Ευρώπης αλλά θα πληρώσουν πολύ ακριβά το τίμημα όσοι κλείνουν τα σύνορα προηγουμένως από τη Γερμανία. Η Γερμανία με τις τράπεζές της ε, προασπίζεται αυτή τη συμφωνία. Και εδώ πρέπει να δούμε ποια είναι τα κριτήρια που θα ε, υπερισχύσουν, θα επικρατήσουν ε, για την διαχείριση των ρόλων των προσφύγων με το σήμα του Ερντογάν, με το σήμα της Τουρκίας. Λέμε για 450.000 που θα φύγουν προς την Ιταλία. Δεν είναι τυχαίο που τα σύνορα κλείνουν από την Τουρκία. Δεν μπορούμε να μην μείνουμε έτσι εκτεθειμένοι στα χέρια ενό τρελού όπω ο Ερντογάν. Εδώ και μέρε η Τουρκία απειλεί να καταγγείλει την ε, συμφωνία. Έχουμε καταγγελίε από τη μεριά τη Διεθνού Αμνηστία. Είναι εξτρεμιστή ο Ερντογάν και λέει ε, ότι ε, εμεί αυτό που θέλουμε είναι ποτέ, ποτέ, ποτέ εισβολή των Τούρκων στην Ευρώπη. Ποτέ, ποτέ. Θα ήθελα να πω στους βουλευτές ότι θα έχουμε πρόβλημα με τη διαδικασία Καξλιά και δεν θα έχουμε χρόνο να μπορέσουμε να δώσουμε σε όλους το λόγο γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο. Μπορείτε να δώσετε την ομιλία σα έγγραφα και ζητώ συγγνώμη γιατί είχαμε αυτά τα προβλήματα. είναι τώρα το λόγο στον κύριο Μπρόκ για 1,5 λεπτό κυρία Πρόεδρε, λέει ο Μπρόκ. Ε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ε, Κομισιόν για το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Αν θέλουμε να έχουμε λιγότεροι πρόσφυγες στην Ευρώπη, αν θέλουμε να έχουμε τα άτομα που έχουν δικαίωμα να έρθουν στην Ευρώπη, αν θέλουμε να καταστήλουμε τη δραστηριότητα των διακινητών και να μην χάσουν πια τη ζωή τους οι άνθρωποι πνιγόμενοι στη θάλασσα, θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία. Είναι απαραίτητο να θυμηθούμε ότι η Τουρκία, ο Λίβανος και η Ορδανία τα τελευταία χρόνια έχουν υποδεχθεί εκατομμύρια ανθρώπους, πολύ περισσότερους από ό,τι εμείς. Είναι καιρός αυτές οι χώρες να ελαφρωθεί το βάρος τους από τους πρόσφυγες γιατί αυτοί είναι, αυτές οι χώρες είναι που είναι υποχρεωμένες να υποστηρίζουν τους πρόσφυγες, να δίνουν τροφή, περίθαλψη και σχολεία στα παιδιά τους. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να σταματήσουν οι άνθρωποι να περνούν τη θάλασσα. Πρέπει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης να βρίσκονται στην Λιβύη, στην Τουρκία. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με θαλάσσια σύνορα, γιατί εκεί οι άνθρωποι βρίσκονται ήδη στη θάλασσα όταν προσπαθούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να μην έχουμε μια Ευρώπη η οποία θα έχει Φράχτε από σηματόπλαμα. Κανεί δεν το θέλει από εμά. κανένα δεν θέλει να το δώσει αυτό ω Ευρώπη στα παιδιά του. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε με του γείτονε μα. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα σταματήσουμε να καταδικάζουμε την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσίων ελευθεριών. Όχι, δεν θα πάρει καμία έκπτωση η Τουρκία για αυτά τα οποία κάνει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί θα υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα λεπτό, η κυρία Ζήπαλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η συμφωνία των χωρών μελών με την Τουρκία δεν είναι η ορθή απάντηση στο προσφυγικό. Ναι, χρειαζόμαστε τη συνεργασία με τρίτε χώρες και με την Τουρκία βεβαίω, Αλλά οι χώρε μέλη δεν, μπορούν να, δεν είναι δυνατόν αναμένουν η Τουρκία να καλύπτει την ε, λυπή αλληλεγγύη εντό τη Ευρώπη, να καλύπτει να την καταστήσει. Και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα σύνορα με τη Συρία, η Τουρκία ε, ανορθώνει ένα τεράστιο και μόνο οι Σύριοι πρόσφυγες ε, έχουν ένα καθεστώς προστασίας. Μία νόμιμη συμφωνία με την Τουρκία θα μπορούσε ενδεχομένως να συμπληρώνει μία κοινή ενδοευρωπαϊκή στρατηγική. Ωστόσο κάτι τέτοιο απουσιάζει. Δεν υπάρχει ούτε μία προστασία των προσφύγων σε όλες τις χώρες μέλη, ούτε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα ευρωπαϊκό ε, επανακατάσταση των προσφύγων, ούτε είναι πρόθυμες χώρες μέλη να δεχθούν τους, προσφύ, τους πρόσφυγες. Ε, οι χώρες μέλη και η Τουρκία θα πρέπει και οι δύο να εργαστούν στην κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φόρντ για ένα λεπτό. Συνάδελφοι, Χάλιβας, στρατηγικό τομέα. Διακυβεύονται θέσει απασχόληση και χρειάζονται επιγόντω ενέργειε. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι και στον αντίκτυπο σε άλλου τομεί. Το αντιτάμπινγκ. είναι πολύ ζωτική σημασία. Το ίδιο και για την, πρέπει να εφαρμοστεί σε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τη μετανάστευση δεν υπάρχει εύκολη λύση. Η συμφωνία με την Τουρκία δεν είναι τέλεια, αλλά μπορεί και να βοηθήσει. Αυτοί που είναι στη ζώνη Σέγγεν ε, χρειάζονται μακροπρόθεσμα πλάνα, σχέδια για να σπάσουν ξεπεράσουν τους δεσμούς με τους διακινητές και να έχουν σωστά προγράμματα διαχείρισης των ε, πυρών. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει την ελεύθερη διακίνηση της υπηκόους τρίτων χωρών για, ως κάποιο είδους ανταμεβή επειδή πέθαναν από κάποιο πόλεμο. Θα πρέπει να πάψουμε να επηρεάζουμε τους, ε, το λαό της Βρετανίας όσον αφορά τον αντίκτυπο των διαπραγματεύσεων με, τους, ε, ε, με την Τουρκία. Οι, οι μετανάστες δεν είναι εγκληματίε, αλλά μπορεί αυτή η κατάσταση να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση από τους τρομοκράτες. Είμαστε σε ένα εγκληματικό κόσμο κόσμο, ζούμε σε έναν εγκληματικό κόσμο και πρέπει να χωνιστούμε κατά αυτού. Καλ Πέλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Πρόεδρε του Συμβουλίου, είναι μια πάρα πολύ συγκινησιακή συζήτηση που κάνουμε σήμερα και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Αν με ρωτήσουν οι ψηφοφόροι μου πόσες φορές έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά, δεν θυμάμαι να απαντήσω. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι απλώς μια συμβιβαστική <clears throat> λύση η οποία θα μπορούσε φυσικά να είναι καλύτερη, αλλά δεδομένων των συγκυριών <clears throat> η απόφαση που ελήφθη είναι η σωστή. Γιατί τη στιγμή που έχει κλείσει ο διάβλος των Δυτικών Βαλκανίων, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να αφήσουμε τους ανθρώπους να δικινούνται χωρίς κανένα έλεγχο. Θα πρέπει να σταματήσουμε το έργο των διακινητών. Ήταν η σωστή απάντηση σε όλα αυτά για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την σταθερότητα και την τάξη στα σύνορα. Ελήφθη λοιπόν αυτή η απόφαση με στόχο να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ζωή 500.000 προσφύγων. Είναι καιρός να βοηθήσουμε την Τουρκία καθώς και τις άλλες γειτονικέ χώρες να αντιμετωπίσουν το βάρος το οποίο επομίζονται. Δεν είναι τέλεια όπως είπα αυτή η συμβαστική λύση η Τουρκία μπορεί να μην είναι σε θέση να τηρήσει απόλυτα τη συμφωνία αυτή. Χρειάζεται λοιπόν έλεγχος και εποπτεία για τα θέματα αυτά. Είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον ο πρόεδρος Ερδογάν για το κατά πόσο θα μπορέσουν να τηρήσουν αυτή τη συμφωνία. Ας δούμε λοιπόν το μέλλον τα hotspots δεν λειτουργούν πολύ καλά, τα συστήματα καταγραφής των προσφύγων θα πρέπει να αναβαθμιστούν, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση των προσφύγων στους καταβλισμούς. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα δούμε γιατί είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ο κ. Μουράης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω συμμερίζομαι πολλέ από τι ανησυχίε σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα που εκφράστηκαν από του συναδέλφου, αλλά α είμαστε ειλικρινεί εδώ σήμερα ότι αυτή η συμφωνία ε, πραγματικά ε, βαρύνει το ζήτημα της ελληνικής. Το πρώτο μου ερώτημα προς την Πρόεδρο είναι το εξής. Εμείς στην Επιτροπή ΛΕΙΜΠΕ, όπου προεδρεύω, ε, συζητήσαμε με τον Μάρτιν Βέρβεϊ και μας απάντησε πολύ ειλικρινά ότι υπάρχουν ε, στα στρατόπεδα και τις διαδικασίες ε, ε, ταυτοποίησης των, των μεταναστών και είπα στο πρόεδρο του Συμβουλίου σε σχέση με την ομιλία που έδωσε στην, αρχή ότι όλοι, όλα, ε, ε, τον ενημέρωση σε σχέση με τα προβλήματα για τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι χώρε μέλη θα παράσχουν του αναγκαίου πόρου, ούτω ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο και να υπάρξουν κάποια εχέγγυα ασφαλεία ότι διαφυλώσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για, ευχαριστώ για 3,5 λεπτά ο κύριος ε, Νίντερμαϊερ κατανοώ απόλυτα τι ανησυχίε όλων αυτών οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προσφυγική κρίση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και το Συμβούλιο για τι ενέργειε τους. Η ταχύτητα των αποτελεσμάτων που επετέθησαν δείχνει πόσο χρόνο χάσαμε πέρσι. Πρέπει τώρα να ατενίσουμε το μέλλον και να εξασφαλίσουμε ότι συνεχίζεται η πρόοδο στην Ελλάδα και να εστιάσουμε σε άλλες περιοχές προβλημάτων για το μεταναστευτικό θέμα όπως πραγματικά χάρη ε, ο διάβλος ε, μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Καλέ και οι άλλες περιοχές της Μεσογείου. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά η εμπειρία μας στην Ελλάδα δείχνει ότι όλα αυτά είναι εφικτά. Να πω κάτι και για την οικονομία. Πριν από λίγες μέρες είπα ότι μου φαίνεται πια ότι τα πολιτικά προγράμματα, πολιτικά προβλήματα είναι πιο μεγάλα από τα οικονομικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, Πρέπει να διατηρήσουμε την πορεία μας για την οικονομική πολιτική. κυβέρνηση. θα πρέπει να τηρήσουν τα συμπεφωνημένα και να βελτιώσουν τη δημοσιονομική τους κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μεγάλη ε, ατζέντα της μεταρρυθμίσης στον φορολογικό τομέα και τις μελλοντικέ συμφωνίες με την Κίνα. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά λοιπόν και για το μέλλον της Ευρώπης και ελπίζω θα τα λάβουμε πολύ στα σοβαρά. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρθία Πέρες, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτή τη ε, συζήτηση περισσεύουν οι βάρες και τις κουβέντες που ορισμένοι χρησιμοποιούνταν μιλώντας για έξοδο, για επιτυχία όταν ε, μιλάμε για τη συμφωνία με την Τουρκία. Ε, καταρχάς όμως θα πρέπει να βάλουμε τάξη στο σπίτι μας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την προφανή αποτυχία της διαχείρισης της ε, μεταναστευτικής κρίσης στους τελευταίους μήνες. Αποτυχία που υποχρέωσε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που ήδη έχει εμφισβητηθεί από ένα μεγάλο αριθμό ανθρωπιστικών οργανώσεων και που τις πρώτες μέρες εφαρμογής της έχει δείξει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και ενώ η κοινή γνώμη μιλά για ντροπή, την ντροπή της Ευρώπης και οι εθνικοί ε, ηγέτες ε, τρίβουν τα χέρια τους, γιατί να μιλάμε για ντροπή της Ευρώπης σημαίνει ότι καλύπτουμε και κρύβουμε την ίδια του στην αντικανότητα να συμφωνήσουν και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που έχουν οι ίδιοι. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στην Ισπανία ε, από πλευρά τη κυβέρνηση του κυρίου Ραχώη έγιναν δεκτοί 18 όλοι και όλοι πρόσφυγες. Πιστεύουμε πραγματικά πως αυτή η ανικανότητα μπορεί να είναι αποδεκτή όταν μιλάμε για τις ζωές δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που φεύγουν από τον πόλεμο και από το θάνατο. Χρειάζεται οι χώρες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, να εφαρμόσουν την αρχή της επικουρικότητας και ε, αυτό γιατί η Ευρώπη διαφορετικά θα κινδυνεύσει. Ας μην γράψουμε την τελευταία σελίδα της ιστορίας μας με, την, ε, ε, με τον πόνο των ανθρώπων. Ο κύριος Ρανζέλ, 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Αυτό το οποίο θα καταστήσω σαφές σε όλους εδώ είναι ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στα πλαίσια της κρίσης των προσφύγων. Να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα των προσφύγων με την υποδοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει αλληλεγγύη και αυτό είναι κεφαλαίωδε. Για να γίνει κάτι τέτοιο, εγώ πιστεύω ότι η συμφωνία με την Τουρκία δεν είναι η καλύτερη συμφωνία, είναι μια συμφωνία εφικτή. Θα πρέπει να είναι η αρχή της δράσης μας για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα των με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ακόμα και εάν υπάρχει ε, επίκριση του Κοινοβουλίου για την πορτογαλική οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Συγχρόνως, όμως, εγώ πρέπει να επενέσω την πορτογαλική κυβέρνηση για τη δράση της υπέρ των προσφύγων. Εμείς ως Πορτογαλία είπαμε ότι όχι μόνο είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε 4.000 πρόσφυγες, αλλά είμαστε σε θέση να δεχτούμε 10.000 ε, πρόσφυγες και έχουμε περάσει τους 1.200 ήδη η Πορτογαλία, η κοινωνία των πολιτών της Πορτογαλίας και η κυβέρνηση της Πορτογαλίας δίνουν ένα καλό παράδειγμα και ελπίζω και οι άλλες χώρες της Ευρώπης να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα γιατί έτσι θα είναι πιο εύκολο να ξεπεράσουμε την κρίση. Ένα λεπτό ο κύριος Βάιντενχολτσα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό ότι αυτή η σύνοδος της τελευταίας στιγμής οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα γιατί καταρχήν η συνεργασία με τη γείτονα Τουρκία, παρόλο που είναι σύνθετη και με κινδύνου, ε, είναι παρέγκλητη. Και ε, είναι σωστά βήματα, θα έπρεπε νωρίτερα να έχουν γίνει έλεγχες στη ζώνη Σέγγεν και θα πρέπει να μεριμνήσουμε να δούμε κατά πόσο όλα εφαρμόζονται σωστά. Πρώτον, η εφαρμογή ε, εμφανίζει κάποιε δυσκολίες γιατί δεν υπάρχει αναγκαίο προσωπικό και υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες που εκφράζονται εκ μέρους ε, των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για συστηματικές παραβιάσεις. Και ε, θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα κατά νου ότι εδώ πρόκειται μόνο για πρώτα βήματα, αλλά χρειαζόμαστε μια, ε, μια μεγάλη μια λύση η οποία θα πρέπει να θέσει ε, στο επίκεντρο της προσοχής της και ως προτεραιότητα το μέλλον των χωρών προέλευσης των προσφύγων. Ευχαριστώ. Κύριος Κάρας. Ευχαριστώ πολύ. Εξάρτημας κυρίες και κύριοι εκφράστηκαν ε, δικαιολογημένα πάρα πολλές ε, ανησυχίες εδώ. Αλλά θα ήθελα εγώ να θέσω το εξής ερώτημα. Διερωτώ με ποια, πώς θα μπορούσε να είχε διαμορφωθεί η παρούσα συζήτηση εάν δεν είχαμε καταλήξει σε μια συμφωνία με την Τουρκία. Εάν η Κομισιόν δεν είχε υποβάλει μια πρόταση για, μια, για τη χάραξη μια κοινή ε, πολιτική ε, ασύλου. Εάν η στρατηγική τη ε, Επιτροπή για ανάπτυξη και απασχόληση δεν είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο γιατί με την αύξηση των εθνικισμών των εγωιστικών τοποθετήσεων της έλλειψης αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα, ε, είχε, θα είχαν οδηγήσει όλα αυτά σε μεγαλύτερη περιχαράκωση των συνόρων και θα μιλούσαν πολύ περισσότερο για μια περιχαράκωση του, της Ευρώπης. Ωστόσο, αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Επιθυμούμε δεν θέλουμε το Μπρένερ να κλείσει. Θέλουμε τα Μπρένερ στην Ευρώπη να παραμείνουν ανοιχτά. Και κυρίες και κύριοι, η συμφωνία αυτή μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον ε, ε, τηρείται το διεθνές δίκαιο και υπάρχει εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόνο εφόσον πραγματικά αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας σε όλες τις χώρες ε, μέλη και εφόσον κατανοήσουμε ότι η συμφωνία με την Τουρκία δεν επιλύει ουσιαστικά το πρόβλημα. Η δομένη εδώ είναι ένα παράδειγμα. Χρειαζόμαστε λύσεις εντός της Ευρώπης και δυστυχώς το Συμβούλιο δεν έφερε αυτές τις ε, λύσεις. Η κυρία Τόρα. Αυτή η συμφωνία προέκυψε από αναγκαιότητα, γιατί ήμασταν με τη θηλιά στο λαιμό, γιατί οι χώρες δεν έκαναν αυτό που έπρεπε η καθεμία. Θα έπρεπε λοιπόν τώρα να επαγρυπνούμε διπλά, να ελέγχουμε τη διαχείριση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Η Ευρώπη είναι υπεύθυνη, δεν μπορούμε να ανύπτουμε τα σχήρα μα έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να δράσει, η Τουρκία πρέπει να δράσει. Όχι, εμεί πρέπει να δράσουμε. Οι ε, γυναίκε και τα παιδιά, τι γίνεται με όλου αυτού φτάνουν ειδήσει ε, για εκμετάλλευση και για ε, υποβαθμισμένε συνθήκε διαβίωση. Αυτό είναι παράδεκτο. Είναι δική μα ευρωπαϊκή ευθύνη, ηθική πάνω απ' όλα και μετά πολιτική και θεσμική. Θέλουμε να, να δούμε αν μπορούν να υπάρξουν hotspot τα οποία θα διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκά. Γιατί μόνο εμεί, άμεσα υπεύθυνοι, θα μπορούμε πραγματικά να επαχρυπνούμε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τέλο, ένα πρόβλημα σταματά και ένα άλλο ξεκινά. Εδώ και λίγε μέρε στην Ιταλία φτάνουν χίλια άνθρωποι την μέρα και για την Ιταλία και για την Μάλτα ήδη από τώρα θα πρέπει να δουλέψουμε με το, υπό, την, υπό το σήμα της αλληλεγγύης και τη Συνεστό. Η κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Σημερινή συζήτηση και η συμφωνία με την Τουρκία ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Αυτή η συμφωνία δεν είναι ιδανική, δεν είναι τέλεια, όπως είπατε και εσείς, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο και απτό βήμα. Όπως είπε ο συναδελφός μου ο κύριος Κάρας, γιατί αλλιώς τι θα συζητούσαμε σήμερα αν δεν είχαμε αυτή τη συμφωνία. Ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν είναι η μόνη λύση για το πρόβλημα αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες με την Τουρκία. Μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα για το αν η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος. Ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί οι μειονότητες και τα μέσα ενημέρωσης αλλά θα πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία και πιστεύω θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αλλιώς αρκετούς ανθρώπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα για να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό ρεύμα και πρέπει να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Είπαμε από την αρχή ότι χρειάζεται αλληλεγγύη και πνεύμα ευθύνη και είναι πραγματικά η δική μα ευθύνη να δώσουμε μια λύση. Έχει κλείσει ο δρόμο των Βαλκανίων και αυτό ήταν μια θετική κίνηση, αλλά αρχίζει και πάλι η ιδίωδος τη Μεσογείου με το να φτιάξουμε φράχτες από σειρματόπλεγμα δεν είναι λύση, τουλάχιστον στη θάλασσα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι η Τουρκία είναι το μόνο η μόνη λύση πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας. Ένα ερώτημα έχω μονάχα για τον κύριο Τάσκ. Πώς θα εποπτεύσετε την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και πώς θα εξασφαλίσετε ότι τα 3 ή 6 δισεκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν σωστά. Η κυρία Βαλεντιάνο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε ε, Επίτροπε, η συμφωνία που έχουμε υπογράψει με την Τουρκία σημαίνει μια μαζική παρέτηση της Ευρώπης από τις ευθύνες που έχουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είναι μια μαζική παρέτηση από τις νομικές μας υποχρεώσεις, από τις πολιτικές μας υποχρεώσεις και από τις ειδικές μας υποχρεώσεις. Εμείς θέλουμε να έχουμε συμφωνήσει με τρίτες χώρες. Ναι, αλλά δεν θέλουμε να αποσύσουμε και να εγκαταλείψουμε τις υποχρεώσεις μας. Τους τελευταίους μήνες, κλείνοντας τα σύνορα, έχουμε δημιουργήσει μια ποντικοπαγίδα για τους πρόσφυγες, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι. Και αφήνουμε την κατάσταση να γίνεται όλο και χειρότερη, να επιδεινώνεται όλο και περισσότερο, χωρίς κανένα έλεγχο. Και αυτό ήταν ακριβώς αυτό το οποίο θέλαν να αποφύγουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ζητώντα από τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν την ευθύνη για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ρευμάτων. Θέλω να μιλήσω ιδιαίτερα για τα παιδιά που δεν τα προστατεύουμε, τα παιδιά των προσφύγων. Είναι αυτά τα παιδιά που χρειάζονται τη μεγαλύτερη προστασία, τα γόρια και τα κορίτσια. Αυτά ξέρετε κύριε Τούσκ ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι απόλυτα παράνομο. Για να μισή λεπτό, ο κύριο Κεφαλογιάννη. Κυρία Πρόεδρε, το να μην υπήρχε συμφωνία στι 18 Μαρτίου θα ήταν μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Όμω τα θετικά σταματούν εδώ η συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας είναι πολύπλοκη σύνθετη ανησυχητικά ασαφής. η συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας μετέτρεψε ένα διεθνές ευρωπαϊκό ζήτημα σε διμερές ζήτημα μεταξύ ελλάδος και τουρκίας. τα ευρωπαϊκά σύνορα έχουν μεταφερθεί στα βόρεια σύνορα της ελλάδος συγκλειδωμένοι τα ελληνικά σύνορα είναι κλειστά. η τουρκία λαμβάνει τρία συν δισεκατομμύρια ευρώ δεν έχει καταπολεμήσει τα κυκλώματα των διακινητών δεν έχει επιβάλει θεώρηση εισόδου στους πολίτες των κρατών από τη βόρεια αφρική που με 30 ευρώ μετακινούνται στην τουρκία και μετά περνούν χωρίς βίζα στα ελληνικά σύνορα και στην ευρωπαϊκή ένωση. δεν έχει υιοθετήσει το πλαίσιο για το άσυλο όπως ορίζεται με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες. η ελλάδα παραμένει εγκλωβισμένη με 53.000 πρόσφυγες η μετεγκατάσταση προσφύγων στις υπόλοιπες χώρες είναι προβληματική και δυστυχώς η μόνη λύση είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η ευρωπαϊκή ακτοφυλακή η διεύρυνση και η εμβάση των δημοκρατικών μας θεσμών. Η, Ελλάδα, η Ευρώπη δείχνει αδυναμία όταν χώρες όπως ο Λίβανος και η Ορδανία μπορούν να υποδέχονται τρία εκατομμύρια πρόσφυγες η Τουρκία το ίδιο και η Ευρώπη δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα εκατομμύριο πρόσφυγες με αξιοπρέπεια όπως τους αξίζει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό για τον κύριο Μαυρίδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι συμφωνούμε πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζονται. Με την Τουρκία αυτό έχει γίνει παράδοση. Και έχει γίνει παράδοση επειδή πηγαίνουμε τουλάχιστον είκοσι χρόνια πίσω η τουρκία δεν εφαρμόζει όλα όσα έχει συμφωνήσει και προσυπογράψει με την ευρωπαϊκή ένωση και αφορούν θέματα βασικών κανόνων δικαίου εντός της ίδιας της τουρκίας αλλά και ειδικότερα σε σχέση με το κράτος μέλος της κυπριακής δημοκρατίας. επομένως αγαπητέ κύριε τούσκ όταν λέμε ότι δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την κύπρο όταν ακούω τον κύριο μπροκ να λέει εμείς θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τουρκία αυτά είναι λόγια. πότε θα αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε τον ερντογάν και να προστατεύσουμε τις αρχές και τους κανόνες δικαίου της ίδιας της ευρωπαϊκής ένωσης. αυτό είναι το ερώτημα. Ένα λεπτό κύριε Ανίμπλα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για να μπορέσουμε να δαμάσουμε και να ελέγξουμε την προσφυγική κρίση, αυτό είναι μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει για την Ευρώπη και η συμφωνία με την Τουρκία είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Δεν είναι επαρκέ από μόνο του, αλλά είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη λύση του προβλήματος αυτό. Γιατί βοηθάει του ανθρώπου να ξεφύγουν από τα νύχια των διακινητών και δίνει και μια συντεταγμένη διαδικασία για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό υποστηρίζω αυτή τη συμφωνία. Βέβαια είναι προβληματικό αυτό το οποίο έχει ε, προτείνει η Τουρκία να δώσει ως αντίτιμο των 6 δισεκατομμύριων ευρώ. Παραμένει το ερώτημα του αν θα πρέπει να ανοίξουμε περισσότερα κεφάλαια από το Συμβούλιο. Εμείς δεν έχουμε εδώ να δώσουμε κάποια απόφαση για το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδίω του κόμματό μου, το οποίο θέλει μια προνομιακή εταιρική σχέση, αλλά όχι την πλήρη ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα θέματα φυσικά θα μα απασχολήσει το Κοινοβούλιο, αλλά έχω ήδη μια πολύ κριτική στάση εναντί τη Τουρκία. Ο κ. Στάνισο, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, Τις τελευταίες ε, εβδομάδες είχαμε πάσες φέσεις ερμηνείες για τη συμφωνία που επετέφθη με την Τουρκία. Ορισμένες αρκετά ακραίες. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεπουληθεί, έχει πουλήσει τη ζωή του στον διάβολο, έχει συνθηκολογήσει κλπ. Ωστόσο ήταν, ε, πρόκειται για μια αναγκαία και χρήσιμη συμφωνία και ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδύναμη και δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει ε, τις ίδιες τις συνθήκες. Και πράγματι ο διάβολος κρύβεται σε λεπτομέρειες. Πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία οικονομικά, γιατί θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες εκεί όπου βρίσκονται. Δηλαδή ε, πιο κοντά στην ε, Συρία, στην Τουρκία, στο Λίβανο και στην Ιορδανία δηλαδή. Δεύτερον, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα εμπόριο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία. Και τρίτον, η συμφωνία αυτή ε, μας έδωσε κάποια ανάσα για να οργανωθούμε αλλά δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει τίποτα άλλο αν δεν χαράξουμε τη δική μας πολιτική. Ε, uh, Έχω κάποια κατανόηση ακόμα και θαυμασμό για τους πρόεδρους Juncker και Τάσκ για τις προσπάθειες να αντιμετωπίσουν αυτή την άνευ προηγουμένου κρίση και δείξανε και ηγετική θέση και θάρρος για να προσπαθήσουν να βρουν λύσεις παρά τις επικρίσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν. Παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο να θεωρηθεί θετική από ανθρωπιστική άποψη αυτή η συμφωνία, είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα εσωτερικά μας σύνορα και να αποτρέψουμε το χάος. Πρέπει όμως να κάνουμε το ίδιο και σε άλλους χώρους αν ο καθένας θα μπορούσε να μιλάει εδώ στο Κοινοβούλιο όποτε θέλει, θα είχαμε χάος. Το ίδιο και με το προσφυγικό ρεύμα. Όπως είπε ο κύριος Γιούνκερ για τα 6 δισεκατομμύρια για την Τουρκία. Δεν πηγαίνουν στην Τουρκία. Πηγαίνουν, πηγαίνουν στους πρόσφυγες για την στέγαση και την παιδεία τους. Και αυτό τα μέσα ενημέρωσης το έχουν ξεχάσει. Και επίσης είπε ο κύριος Γιούγκερ, ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να βοηθούμε και τους ανθρώπους που είναι ήδη στην Ευρώπη πρόσφυγες. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Ζουρίνιου. Ε. Βόντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, το Συμβούλιο ανέκρινε μέσω της συμφωνίας με την Τουρκία και την ε, επιβεβαίωση των προτεραιοτήτων της πολιτικής άμυνας και κοινή ε, άμυνας και ε, ασφάλειας σε μία λύση για την κρίση της, των προσφύγων. Όμως, ενέκρινε και την ε, συνέχιση των ε, ε, δημοσιονομικών πολιτικών και επίσης συμφώνησε, δεσμεύθηκε τον Ιούνιο να δώσει μια νέα όθηση στην ενιαία αγορά, στην ψηφιακή αγορά, αλλά και στην Ένωση των Κεφαλαγορών. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση μόνο έχει νόημα. Τι περιμένουν τα κράτη-μέλη για να αρχίσουν να εφαρμόζουν αυτά που τα ίδια ενέκριναν Φτάνουν τα λόγια, χρειαζόμαστε καλά παραδείγματα. Η Πορτογαλία δεν περιμένει, δρά. Ε, ε υποδέχεται το διπλό άσιο των προσφύγων που είχαν συμφωνηθεί αρχικά και προχωρά σε ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ανάπτυξη που έχει. Χρειαζόμαστε λοιπόν δράσει, ε, καλά παραδείγματα που θα πολλαπλασιαστούν. Ευχαριστώ. Κύριο Χόκουμαρκ, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, δύο συμπεράσματα για όσους ε, θέλουν να διχάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να, να την κατακαιρματίσουν. Η πρόκληση του μεταναστευτικού είναι μακροπρόθεσμη. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις για το πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να είμαστε επικριτικοί απέναντι στι διάφορες λύσεις, ίσως γιατί καμιά λύση δεν θα ήταν τέλεια ούτως ή άλλως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αν δεν δράσουμε από κοινού, δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν θα μπορέσουμε καθόλου να δράσουμε. Και αυτό θα ήταν κρίμα απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεφεύγουν από βιαιότητα, από φρικαλαιότητες. Και αυτό θα ήταν μια ντροπή που θα μας βαρύνει θα βαρύνει όσους θέλουν να διχαστούμε και να μην μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας. Δεύτερον, Ουκρανία. Αν στρέψουμε τα νότα μας στην Ουκρανία, αφήνουμε ελεύθερες τις δυνάμεις τους κότους που υπονομεύουν την ευρωπαϊκή σταθερότητα και αυτό είναι ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Στηρίξτε την Ουκρανία. Διασφαλίστε τους ότι μπορούμε να σταθούμε ως Ενωμένη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο κύριος Ανδρουλάκης. Ένα μήνα πριν, στη συζήτηση για την επικείμενη συμφωνία, σας προειδοποιούσαμε για τα νομικά κενά. Εσείς όμως δώσατε στον κύριο Ερντογάν τη δυνατότητα να λειτουργεί εκβιαστικά και να απαιτεί όλο και μεγαλύτερα ανταλλάγματα για να κάνει το αυτονόητο. εάν πράγματι είναι τόσο ασφαλή χώρα η τουρκία γιατί δεν ζητάμε τον κύριο μπέρνεμαν που τόσο ενόξε το πείμα του τον κύριο ερντογάν να το απαγγείλει στην άγκυρα ή την κωνσταντινούπολη. σήμερα τρει εβδομάδε μετά την έναρξη τη εφαρμογή α είμαστε ειλικρινεί οι ροέ έχουν μειωθεί όχι γιατί λειτουργεί η συμφωνία αυτή καθεαυτή αλλά γιατί έχουν κλείσει τα βόρεια σύνορα τη εφαρμογη α ειμαστε ειλικρινει οι ροε εχουν μειωθει οχι γιατι λειτουργει η συμφωνια αυτη καθεαυτη αλλα γιατι εχουν κλεισει τα βορεια συνορα τη ελλαδο κάποιοι βολεύονται με την κατάσταση καθώς πλέον δεν φτάνουν πρόσφυγες στα σύνορά τους. γι' αυτό κάνουν πως δεν βλέπουν πως η ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια αποθήκη ψυχών με εικόνες σε ειδωμένη και πειραιά που δεν τιμούν τις ευρωπαϊκές αξίες. αν θέλουμε λοιπόν να εκπροσωπούμε το όραμα της ενωμένης ΕΕ, το όραμα της αλληλεγγύης πρέπει να επιβάλλουμε τη διαδικασία της μετεγκατάστασης. και αν κάποιοι δεν θέλουν να υλοποιήσουν γιατί έμαθαν να παίρνουν από την ευρώπη ότι τους βολεύει ή γιατί χρησιμοποιούν τον εθνολαϊκισμό ω όπλο εσωτερική κατανάλωση τότε να έχουν ανάλογε κυρώσει με περικοπέ των διαρθρωτικών ταμείων. Κύριε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το θέμα της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έχουν λεχθεί περίπου όλα. Απλώς θα ήθελα να δείξω δύο ακόμα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το πρώτο είναι αυτό που λέει ότι τον Ιούνιο στην ε, σύνοδο της 28ης Ιουνίου θα εξεταστεί το θέμα της ε, συμπλήρωσης της ε, ενιαίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο που θέλουμε ο Βρετανικός λαός να πει ναι στη συμφωνία η οποία επετέφθη ανεξάρτητα λοιπόν από αυτό το αποτέλεσμα εμείς θα πρέπει αμέσως να θέσουμε επιτάπητο στο θέμα της ε, συμπλήρωσης οικονομικής και νομισματικής ένωσης, γιατί αυτό το θέμα έχει χρονίσει πάρα πολύ. Είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να εδραιώσουμε αυτό το βασικό υπόβαθρο της Ευρώπης. Μετά έχουμε το θέμα της χαλιβουργίας. Ευτυχώς οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έκρουσαν το κόνδυνα του κινδύνου. Υπάρχει υπερπαραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό οδηγεί σε προβλήματα στη χαλιβουργία της στην Ευρώπη πρέπει η Ολλανδική Προεδρία να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για εμπορική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δοθούν απαντήσεις γιατί αυτό περιμένουν από την Κομισιόν οι Ευρωπαίοι. Ο κύριος Μάμικινς για ένα μισή λεπτό. Κύριε Τούσκ, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ υποστηρίζω μια επικοδομητική σχέση με την Τουρκία. Αλλά η τωρινή σχέση μάλλον θυμίζει μια σχέση εκβιασμού από τον πρόεδρο Έρντογαν ο οποίος είναι έτοιμος να πλημμυρίσει την Ευρώπη με προσφύγες αν δεν υποκύψει η Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει επίσης και με το, την ε, θέληση της Τουρκίας να υπάρχει ίσως στην Ευρώπη χωρίς ε, βίζα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια. Αλλά η στάση της Τουρκίας έναντι της Ευρώπης δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως είναι. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η Τουρκία παίζει σημαντικό ρόλο στο να ενισχύσει ε, ομάδε ομάδες όπως το Ισλαμικό κράτος και η Τζαμπάτ Αλνούσρα στη Συρία. Αυτό έχει οξύνει την κρίση και των προσφύγων. Ζητώ από τους Ευρωπαίους ηγέτες να ενισχύσουν και να προωθήσουν το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το να παραμείνουν πιστοί στις αξίες μας. Ευχαριστώ. Προσκαλώ τώρα τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο να απαντήσει και σας δίνω το λόγο. E, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Τούσκ. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ε, ουσιαστικές σας ε, συμβολές, πολλές εκ των οποίων είναι ευθυγραμμισμένες με τους στόχους και τις ιδέες της Επιτροπής. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια στοιχεία. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι ανταγωνιστικές όσον αφορά ε, δυνάμεις ε, ε, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα με κοινό τρόπο η, η Ευρώπη και η Τουρκία είναι υπό μεγάλη πίεση αντιμετωπίζουν το, τις ίδιες προκλήσεις και αν προηγουμένου κατάσταση η συνεργασία είναι απαραίτητη είναι αλήθεια ότι η Τουρκία θεωρεί αυτή τη συνεργασία ως καταλήτη για να αναζωογονήσει τις σχέσεις μας καθώς και την ευρωπαϊκή της προοπτική. Ε, αυτό το νέο κεφάλαιο δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ωστόσο ως υποχώρηση απέναντι στις βασικές αρχές και αξίες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αντιθέτως, πρόκειται για μια ευκαιρία για την Τουρκία να έρθει πιο κοντά στα ευρωπαϊκά στάνταρ, ευρωπαϊκά προδια, ευρωπαϊκές προδιαγραφές, δημοκρατικές αξίες, κράτος δικαίου, ελεύθερη έκφραση, σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και επίλυση του Κυπριακού. Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να υπάρχει, ε, να είναι γείτονά μας μια δημοκρατική και σταθερή Ευρώπη και είναι στο συμφέρον της Τουρκίας να έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση σταθερό υποστηριχτή και εταίρο. Η προσφυγική κρίση μας έφερε πιο στενά ε, σε ένα πνεύμα κοινή συνεννόησης. Το θέμα είναι να δείξουμε αν εννοούμε αυτό που λέμε και αυτά που συμφωνούμε. Παρακολουθούμε έτσι ώστε οποιαδήποτε πτυχή αυτής της συμφωνίας να υλοποιηθεί σε πλήρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Ε, δεν υπάρχει αμφιβολία καμία περί αυτού. Για παράδειγμα, οι τουρκικές αρχές έχουν περάσει νομοθεσίες για να εξασφαλίσουν την προστασία των σύρων. Είμαστε πολύ ρητά τους είπαμε ότι χρειάζονται εγγυήσει για όλους όσοι χρειάζονται προστασία. ΣΥΡΙ ή μη ΣΥΡΙ. Για την απελευθέρωση των θεωρήσεων ε, έχουμε, ε, ε, θα απαιτούμε 72 προαπαιτούμενα, αλλά η Κομισιόν ήταν ξεκάθαρη. η μόνη πρόταση για άρση των θεωρήσεων αν τηρηθούν όλα τα ορόσημα και η, γνω... η... η Τουρκία το γνωρίζει αυτό και καταβάλει προσπάθειες για να μπορέσουμε να άρουμε μέχρι τον Ιούνιο του 2016 τις θεωρήσεις. Η συμφωνία μόλις άρχισε να, να εφαρμόζεται, 300 άνθρωποι έχουν επιστραφεί που δεν ζήτησαν άσυλο και 74 ε, Σύριοι έχουν φύγει ε, ε, από την Τουρκία κατευθείαν. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Την επόμενη εβδομάδα η Κομισιόν επισήμως θα κάνει αναφορά για την εφαρμογή όλων των βημάτων αυτής της συμφωνίας. Θα σας πω όμως το εξής. Αυτή η συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα για μια μακροχρόνια σχέση. Κοινό στόχος είναι να έρθουμε πιο κοντά μεν στους δε όσον αφορά τις αξίες όπως τόνισα στην αρχή το εισηγησής μου. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν ε, στην Ελλάδα ε, βρίσκεται παντού, κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την Ελλάδα να επεκτείνει τις δυνατότητές της, τη χωρητικότητα, έτσι ώστε ευάλωτοι ετούντες όπως οι γυναίκες και παιδιά να έχουν τη σωστή μεταχείριση. Οι άνθρωποι μας είναι εκεί ε, σε όλα τα ελληνικά νησιά αλλά και στην ενδοχώρα και παρέχουμε τη βοήθειά μας προς την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές. Τα κράτη-μέλη χρειάζεται να συνεχίσουν να επαναγκαθιστούν μασικά από την Ελλάδα και ε, επιμένω σε αυτό ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να, λάβουν το μερίδιο, να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης τους. Πάνω από 50.000 άνθρωποι έχουν κολλήσει στην Ελλάδα το 70% τουλάχιστον εξ αυτών είναι επιλέξιμοι για επανεγκατάσταση. Αυτοί που βρίσκονται στην Ιδωμένη και στον Πειραιά ε, ήδη πριν τις 20 Μαρτίου βρίσκονταν εκεί. Οι αφήξει τώρα από την Λιβύη στην Ιταλία δείχνουν ότι από τη στιγμή που επικρατεί αστάθεια, που υπάρχουν διακινητέ που εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, ο κόσμο θα συνεχίσει να μεταναστεύει. Είναι απλούστατο. Πρέπει να δουλέψουμε ε, λοιπόν ευρύτερα, έχοντα την ευρύτερη εικόνα στο μυαλό μα. Δηλαδή, να, να συνεχίσουμε τι προσπάθειε για να επανέλθει η σταθερότητα στη Συρία και στη Λιβύη και άρα να υλοποιηθούν οι πρότασή μα για συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή ευρωπαϊκού επίπεδου. Είμαστε ευτυχεί που το Κοινοβούλιο υπέβαλε έκθεση με χρονοδιάγραμμα που αντικατοπτρίζει αυτέ τι δεσμεύσει. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο εδώ. Μάλιστα το καλοκαίρι έχει και όλα φτάσει. Αυτό σημαίνει αύξηση νομίμων διόδων για τους ανθρώπους, ώστε να μην πρέπει να καταφεύγουν στις στην παράνομη είσοδο. Και θέλω να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές που το ε, ε, ε, που το αυτό το θέμα και το υποστηρίζουν. Ε, πρέπει να παίξουμε Λίβανος, Τουρκία και Ιορδανία έχουν δεχτεί τεράστια πλήθη προσφύγων. Αν θέλουμε όμως να ρυθμίσουμε το πρόβλημα μιας και διαπαντός πρέπει να ανοίξουμε ένα ασφαλές και νόμιμο παράθυρο. Η Ευρώπη χειρό ούτε είναι επιθυμητή ούτε είναι και εφικτή. Ακριβώς επειδή ο κόσμος πάντα θα έχει λόγος για να φεύγει να μετακινείται και να συνεχίζει να προσπαθεί να φτάσει στην Ευρώπη. Όχι μόνο ηθικών, ηθική και νομική ευθύνη να προσφέρουμε ασφάλεια σε όσους το χρειάζονται, αλλά πρέπει να δούμε και τις πολιτικές μας για, την, μελλοντική μας πολιτική. Η μετεγκατάσταση είναι η νόμιμη ε, λύση για όσους χρειάζονται προστασία. Ορισμένοι ανέφεραν το Δουβλίνο. Δεν θέλουμε μια ε, καλολογική μεταρρύθμιση. Θέλουμε ε, μια βαθιά μεταρρύθμιση και βελτίωση του Δουβλίνου ώστε να εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη και την ενσωμάτωση στο νέο σύστημα γιατί αυτό το σύστημα δεν ε, μπορεί να επιβιώσει. Γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όμως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε και όχι ε, να αντιπαλεύουμε ένα στον άλλον. Αυτό ισχύει για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη, αλλά και τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας. Ευχαριστώ. thank you, Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Συμβουλίου θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη που βρίσκονται στους διαδρόμους παρακαλώ να ε, παρακολουθήσουν, να, έρθουν, να, θέσεις και να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση. Κύριε Τούσκ, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν διάφορα, διάφορες πτυχές στη συζήτηση στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Καταρχήν η επανεγκατάσταση. Η επανεγκατάσταση ε, θα αποτελέσει ένα από τα στοιχεία κλειδιά της ευρωπαϊκής ε, λύσης στο προσφυγικό. Και ε, βεβαίω υπό την έννοια αυτή χρειαζόμαστε απαραίτητο ένα πνεύμα αλληλεγγύη. Αλλά θα ήταν ένα σφάλμα εάν θεωρούσαμε ότι είναι το βασικό εργαλείο της πολιτικής μας. Γιατί είναι ένα απλό κίνητρο για την περαιτέρω διαχείριση των μεταναστευτικών ροών όχι ενθάρρυνση νέων ε, προσφυγικών ροών. Δεν είναι αυτό που επιθυμούμε. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να περάσει ξεκάθαρα προς τα έξω σαν μήνυμα. Ε, στην παρούσα συζήτηση ε, ο κ. Φερχοστάτ αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία εν σχέση με την παράτυπη μετανάστευση όσον αφορά τις οδούς της ε, Μεσογείου. Ε, και πραγματικά είμαι πολύ προσεκτικός όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα. Αλλά σήμερα πράγματι αξίζει να τα εξετάσουμε, να αξιολογήσουμε αυτά τα στοιχεία. Γιατί όσον αφορά τη Βαλκανική Οδό είναι αλήθεια ότι 150.000 ε, παράτυποι μετανάστες έφτασαν στην Ευρώπη από την αρχή αυτού του έτους. Αλλά οι, αριθμοί αυτοί μειώνονται μήνα ανά μήνα. Από 70.000 τον Ιανουάριο σε 50.000 τον Φεβρουάριο και 30.000 τον Μάρτιο και είναι περίπου, ήταν περίπου χίλιοι τον Απρίλιο. Ε, φανταστείτε λοιπόν, εάν μόνο το μήνα Ιανουάριο ε, μεσούντος του χειμώνος ε, ήταν 70.000 μετανάστες πόσοι θα έφταναν ε, στην Ευρώπη τον Απρίλιο εάν ε, δεν είχαμε αναλάβει δράση. Δεύτερον, είναι επίσης αληθές ε, ότι από την αρχή αυτού του έτους 20.000 παράτυποι μετανάστες ήρθαν στην Ευρώπη μέσω της διόδου της κεντρικής Μεσογείου και έκτοτε οι αριθμοί πέφτουν. Αλλά μεταξύ αυτών δεν συγκαταλέγονται Σύριοι. Υπάρχουν άλλες εθνικότητες ε, από αφρικανικές χώρες, από την Ιγυρία, από τη Σομαλία, από τη Γάμπια, από τη Γουινέα, Δημοκρατία της Γουινέας και την ακτή του Λεφαντοστού. Τι σημαίνει αυτό, τι θα σήμαινε εάν δεν είχαμε κλείσει την διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτή τη στιγμή θα είχαμε τρεις, ε, τριπλάσιους πενταπλάσιους ε, μετανάστες τόσο από την Αφρική μέσω της Λιβύης καθώς και εκείνους ε, που αυτή τη στιγμή έχουν αναχαιτιστεί ή μάλλον έχουν σταματήσει ή έχουν, στα σύνορα έχουν αποθαρρυνθεί στο να διασχίσουν τα σύνορα. Πολλοί είπαν σήμερα ότι η προτεραιότητά μας θα ήταν να συστήσουμε μια ευρωπαϊκή εκτοφυλακή. Εγώ είμαι υπέρ αυτού, έστω και αν αυτή η εκτοφυλακή δεν θα μπορεί να είναι λειτουργική κατά τη διάρκεια αυτού του έτου. Αυτό είναι αδύνατο. Αλλά θα πρέπει να διορτηθούμε το εξή. Τι θα έπρεπε, έπρεπε ακριβώς να κάνει αυτή η Ευρωπαϊκή Εκτοφυλακή να επιτρέψει την είσοδο σε όλου όσου επιθυμούν να έρθουν στην Ευρώπη ή να του σταματήσει και να του ελέγξει. Η απάντηση νομίζω ότι είναι προφανή ότι θα πρέπει να του σταματήσει και να του ελέγξει το οποίο σημαίνει ε, επίσης μια ε, ισοδυναμία με, την αντιφατική ακριβώς ε, δράση, το αντιφατικό μοντέλο το οποίο εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή. Και καταρχήν θα πρέπει να περιμένουμε από τις εθνικές ακτοφυλακές να εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο στα ευρωπαϊκά σύνορα. Η ευρωπαϊκή ακτοφυλακή θα πρέπει να υποστηρίζει αυτούς οποίους χρειάζονται βοήθεια, αλλά δεν είναι δυνατόν να τις αντικαταστήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πρόεδρε κύριε Τούσκ Και ευχαριστούμε συνάδελφοι. Αυτή η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί και θα ήθελα να πληροφορήσω το σώμα ότι πριν περάσουμε στην επίσημη πανηγυρική συνεδρία με τον πρόεδρο της Πορτογαλίας, κύριε Φερχόφστατ, με συγχωρείτε, προσπαθώ να κάνω μια αναγγελία. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πληροφορήσω το σώμα ότι πριν από την επίσημη συνεδρίαση με τον πρόεδρο της Πορτογαλίας ε, θα έχουμε τα τρία θεσμικά όργανα τα οποία θα υπογράψουν